ξεκινήσουμε πολύ σύντομα. Και να καλωσορίσω την κυρία Σεσίλια Μάλμστρομ, που έχει οριστεί επίτροπος για θέματα εσωτερικά. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Αποτελεί τιμή για μένα ευκαιρία που έχω να καλωσορίζω εδώ την κυρία Μάλπστρομ ως υποψήφια επίτροπο στο σημαντικό χαρτοφυλάκι όπου της ανατέθηκε στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος για το τομέα των ιστορικών υποθέσεων. Η παρούσα ακρόαση θα διαρκέσει τρεις ώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και πάλι να προσέξουμε την πειθαρχία στη διαχείριση του χρόνου σε όλες μας τις παρεμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε λάβει από την Επιτροπή Απασχόληση και από την Επιτροπή Γυναικών ε, κάποια αιτήματα, θα γίνουν τρεις ερωτήσεις από τους τομείς αυτούς και τρεις από την κάθε μια επιτροπή δηλαδή, και συμφωνήσαμε με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων έτσι ώστε οι 27 συνολικά ερωτήσεις που θα γίνουν ε, στην Επίτροπο, την υποψήφια Επίτροπο, θα έχουν για κάθε ερώτηση οι ομιλητές ακριβώς ένα λεπτό. Και η υποψήφια Επίτροπος θα απαντά ε, στην κάθε ερώτηση δύο λεπτά. Θα ακολουθεί συμπληρωματική ερώτηση. De la primera, con una nueva oportunidad por parte de la... Και ε, θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια και πάλι η υποψήφια επίτροπο, να απαντά ένα λεπτό αυτή τη φορά στη συμπληρωματική ερώτηση. Έτσι, ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση, ένα λεπτό συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό δευτερολογία τη ε, υποψηφίας επιτρόπου, η απάντηση δηλαδή. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους βουλευτές, συναδέλφους, να τηρούν το χρόνο τους, 27 που θα ερωτήσουν, για να μην με υποχρεώσετε να σας διακόψω και να μπορούμε με ευελιξία να χειριζόμαστε το χρόνο όπως άλλωστε πράξαμε και στην ακρόαση της υποψηφία Επιτρόπου κυρίας Ρέντινγκ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και παρακαλώ την υποψήφια να σεβαστεί και το δικό της χρόνο και στην αρχική της παρουσίαση και στην έκθεση του προγράμματός της, τα δέκα λεπτά που έχει στη διάθεσή της. Ελπίζω να είναι αγαστή συνεργασία, το ευχόμαστε, ε, μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κρίσιμη η καιρή, ε, συμπίπτουν με τη θέση σε ισχύ της Σύνθεξης Λισαβόνας και αναδύεται το σημαντικό κεφάλαιο εκεί, ο χώρος ελευθερίας ασφάλεια και δικαιοσύνη, το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη και η θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Χάρτη ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Καλώ όρισατε και πάλι, κυρία Μάλστρομ, Έχετε μέσα στο λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ε, Κύριε και κυρίες βουλευτές της Επιτροπής, ε, είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ εδώ σήμερα ως ε, Επίτροπος που έχει οριστεί για θέματα ε, εσωτερικών υποθέσεων. Πολλοί από εσά θα με γνωρίζετε από την θητεία μου ως Ευρωβουλευτή ή από τις πολλές συζητήσεις που είχαμε το φθινόπορο εδώ στο Κοινοβούλιο σας επί Σουηδικής Προεδρίας. Τώρα βρίσκομαι εδώ απέναντί σα ε, και ε, προσλέπω σε μια θετική συνεργασία τα επόμενα πέντε χρόνια. Το Δεκέμβριο υιοθετήθηκε το πρόγραμμα Στοχόλμη ε, και ταυτόχρονα τέθηκε σε ισχύ και η συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτά και τα δύο γεγονότα επηρεάζουν τι επηρεάζουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και με το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης ε, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να ε, ασχοληθούμε με θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το εργανομένο έγκλημα ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αυξανόμενης μετανάστευσης και πρόκειται για τομείς όπου υπάρχει σαφής ε, προστιθέμενη αξία ε, σε μια συνεργασία στα πλαίσια της Ευρώπης. Επίσης γνωρίζω ότι εμείς ως εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, έλλειψης νομιμότητας. Φυσικά μας ανησυχεί το ότι πέφτει το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Ε, μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ακούγοντας ε, τι θέλουν οι άνθρωποι, τι επιθυμούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρουσιάσουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερο διάλογο με το κοινό και την κοινωνία των πολιτών και να εξηγήσουμε τι κάνουμε και γιατί. Η ευθύνη αυτή ε, βρίσκεται στους ώμους όλων μας εδώ μέσα. Ε, το πρόγραμμα Στοκχόλμης μας δίνει τη δυνατότητα ε, να φροντίσουμε οι ανησυχίες των πολιτών να βρίσκονται στο, κέντρο, στο επίκεντρο των εργασιών μας. Και τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω τα έχω πάρει από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. και στην στο προτεραιότητας ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου του Νοεμβρίου. Ε, θέλω να υπερασπιστώ τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλη η συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στις ε, κοινέ μας αξίες, ε, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές χωρίς εξαιρέσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ζουν σε μια ασφαλή Ευρώπη όπου η όπου θα εγγυόμεθα την ασφάλεια τους και την νομική ασφάλεια. Η αλληλεγγύη θα είναι λέξη κλειδί για μένα και μιλάω για αλληλεγγύη ανάμεσα στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτό κατά την, ε, ε, κατά την αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημιουργίας ενός ε, συστήματος ε, ασύλου και μετανάστευσης. Πρόκειται για αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλες τις αρχές καταπολέμησης του εγκλήματος που θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, που έχουμε μπροστά μας και πρόκειται για αλληλεγγύη ε, εντός της ε, Κομισιόν. Να γίνω τώρα πιο συγκεκριμένη. Καταρχήν, θέλω να αναπτύξω μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Μια σφαιρική προσέγγιση, συνεργασία με τρίτες χώρες θα παρέχει ασφάλεια στους σε αυτούς, προστασία σε αυτούς που την χρειάζονται, ε, θα προωθήσει την ε, νόμιμη μετανάστευση και ε, θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε την λάθρομετανάστευση. Η πολιτική ασύλου είναι η δυνατότητα να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται τις αξίες της. Γι' αυτό θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια περιοχή προστασίας αυτών που διώκονται και θα πρέπει να υπάρχει ε, αλληλεγγύη, προβλεψιμότητα και ε, μοίρασμα των ευθυνών και θα πρέπει να ε, σεβαστούμε την συνθήκη της Γενέβης και την αρχή της μη επαναπροώθησης. Με μια τέτοια πολιτική μια τέτοια πολιτική μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνο εάν ασχοληθούμε και με τη λαθρομετανάστευση ταυτόχρονα και αποτελεσματικά. Ε, έχουμε την εσωτερική αγορά που σημαίνει ότι οι πολίτε μα μπορούν να ε, κινούνται ελεύθερα στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή δεν έχουμε εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να ελέγξουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μα σύνορα. Και ε, εδώ εμπίπτει μια πολιτική επανεισδοχής η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης θέλω να δημιουργήσω ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, έχουν πληθυσμό που γυράσκει και ε, χρειάζεται μια δυναμική και ευέλικτη αγορά εργασίας. Φυσικά η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αλλά στο μέλλον θα χρειαστεί να αυξήσουμε την μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς την Ευρώπη. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω τα ε, πλεονεκτήματα του να φτάσει κανείς στην Ευρώπη με νόμιμο και ρυθμισμένο τρόπο. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μια ε, κατάσταση η οποία, ε, από την οποία να μπορούν να κερδίσουν όλοι. Δηλαδή να έχουμε ε, καλές συνθήκες εργασίας και να αναπτύσσεται ταυτόχρονα η κοινωνία της Ευρώπης. Επίσης θα χρειαστούμε καλύτερη πολιτική ένταξη ώστε οι μετανάστες να λειτουργούν σωστά ε, στην κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας μετανάστευσης ε, που θα προστατεύει τα ε, δικαιώματα των μεταναστών με τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θέλω να κάνω μια επισκόπηση όλη τη νομοθεσία και πολιτική στον τομέα για να βελτιώσω το συντονισμό στον τομέα αυτών. Επίση, θέλω μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας η οποία θα πρέπει να μας καταστήσει ικανού να εκμεταλλευτούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ε, απειλές, ε, να υπερασπιστούμε την ελευθερία και τα δικαιώματα. Και είναι σημαντικό να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι ε, στα σοβαρά προτιθέμεθα να αντιμετωπίσουμε την, ε, το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, ε, την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, την παιδική πορνογραφία, την ε, διαφθορά, το κυβερνοέγκλημα και τα ναρκωτικά. Η Frontex, η Europol και η SEPOL έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν εδώ και επίσης θα πρέπει να ε, εμβαθύνουμε συνεργασία με τη Eurojust και την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, θα ξεκινήσω λοιπόν από τη Frontex. Αποτελεσματική συνεργασία προϋποθέτει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και στόχος μου είναι αυτό να γίνει με υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών ε, δεδομένων. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ισχυρός εταίρος σε έναν ε, όλο και πιο παγκοσμοποιημένο κόσμο. Η... Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τους γειτόνους μας ε, και τους εταίρους μας ε, Και ε, ένα από τα πρώτα μέτρα μου ως ε, επίτροπος θα είναι να παρουσιάσω ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοχόλμης. Αυτό θα το κάνω σε συνεργασία με την Βιβιάν Ε, Το πρόγραμμα αυτό θα βασίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις. Και τώρα που ε, έχει υιοθετηθεί το πρόγραμμα της Στοχόλμης όλες οι αποφάσεις μου σχεδόν ε, θα ε, λαμβάνονται ε, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό βρίσκω ότι είναι θετικό και σημαίνει ότι θα συνεργαστούμε στενά εγώ και εσείς τα επόμενα πέντε χρόνια. Όσον αφορά την διαφάνεια, θα φροντίσω εσείς και το Συμβούλιο να λαμβάνετε τις ίδιες πληροφορίες σε όλα τα θέματα. Θέλουμε καλύτερη νομοθεσία και οι προτάσεις της Κομισιόν να είναι πιο ευκολονόητες. Κύριε Πρόεδρε, έχω πολύ σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχω γνωρίσει από μέσα. Ξέρω πόση αφοσίεση και πόση και πόση γνώση υπάρχει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που να είναι ασφαλής, όπου να υπερσπιζόμαστε τα ε, δικαιώματά μας σε μια Ευρώπη η οποία να ασχολείται με τα προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους. Ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, να ε, παρέχουμε μια ανθρώπινη και δίκαιη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης και που προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα κατάσταση μεταναστευση. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να παρουσιάσω αποτελέσματα σε αυτούς του σημαντικούς τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Μάλτρον. Επιταχύνετε για να τηρήσετε το δεκάλεπτό σας, είναι ένα λεπτό επί Ελπίζω να παραμείνουμε στο χρονοδιάγραμμά μας και να το τηρήσουμε. Αρχίζει ο χρόνος των ε, ερωτήσεων σύμφωνα με το σύστημα αντεχόντ και το κανονισμό μας. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Σάιμον Μπουσουτήλ. Um Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε κύματα λαθρομεταναστών από τις αφρικανικές ακτές να φτάνουν στην Ευρώπη. Οργανωμένο έγκλημα προωθεί αυτή τη σκανδαλώδη κατάσταση στον 21ο αιώνα. Είναι ε, ανθρώπινες τραγωδίες αυτές. Εκατοντάδες συνάνθρωποι μας πνίγονται στις θάλασσές μας κάθε χρόνο. Και αυτό επιβαρύνει άλλωστε και δυσανάλογα τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να διασώζουν τους ανθρώπους αυτούς, να τους ε, υποδέχονται και να τους ε, περιθάλπουν. Οι λαοί των χωρών αυτών σήμερα παρακολουθούν την ακρόασή σας και θέλουν να ακούσουν μια σαφή δέσμευση για να σταματήσει ε, διαπαντός αυτή η κατάσταση. Έχω λοιπόν απλή ερώτηση. Θα δεσμευτείτε προς την κατεύθυνση αυτή, θα σταματήσετε για πάντα την λαθρομετανάστευση και πώς θα το κάνετε αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάστρομ. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Συμφωνώ ότι λαμβάνουν χώρα στη Μεσόγειο πραγματικές τραγωδίες και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Η Ευρώπη έχει ευθεία, ευθύνη να λάβει και να δώσει ε, καταφύγιο σε όσους χρήσουν προστασίας με βάση τη συνθήκη της Γενέβης ε, στα πλαίσια του ασύλου και της ε, πολιτικής ε, μη επαναπρόθεση. Αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη λαθρομετανάσταση παρόλα αυτά και το οργανωμένο ε, έγκλημα, το λαθρεμπόριο και τη διακίνηση προσώπων. Δεν ξέρω αν μπορώ μόνη μου να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, αλλά είμαι πρόθυμη να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη Frontex, όπω είπα και στην εισαγωγή μου, θα την ενισχύσουμε αυτή την υπηρεσία, θα αυξήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ούτω ώστε να υπάρχει επιμερισμό πραγματικό των ευθυνών και πολύ σύντομα θα έχουμε ε, το γραφείο του ασύλου στη Μάλτα, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει για να διευκολύνει την κατάσταση. Επίσης, Έχουμε προγράμματα επανεγκατάστασης ε, τα οποία θα επαναξιολογήσουμε και ίσως ε, τα καταστήσουμε έτσι πιο μόνιμα. Θα το δω όταν θα έχουμε έτοιμη την αξιολόγηση. Και φυσικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες για να δούμε πώς μπορούμε ε, με τις όμορες χώρες ε, γύρω από τη Μεσόγειο, με τις χώρες ε, διέλευσης να συνεργαστούμε και να εμπλακούν και αυτές οι χώρες ώστε να σταματήσει αυτή η ηλεκτρομετανάστευση. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια δράση. Από την εποχή του Αδάν και της Εύας και από την εποχή που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών υπάρχουν διαφορές πολιτικές, οικονομικές κτλ. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική που να έχει μια εξωτερική διάσταση για να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις χώρες. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα περίπλοκο θέμα και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο και μαζί σας προκειμένου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ο κ. Μπουσουτήλη για μια δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ. Ε, πρέπει να ευχηθούμε ότι θα γίνει κάτι αυτό που είπατε. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα πρέπει υποτίθεται να βοηθήσει τις ε, χώρες της Νοτιάς Ευρώπης για να βοηθήσουν τους ε, μετανάστες που φτάνουν ε, στην επικράτειά τους και να υποφελθεί και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. αλλά θέλουμε ουσιαστική αλληλεγγύη, όχι αλληλεγγύη στα λόγια. Θα ήθελα να μου πείτε ε, με περισσότερε λεπτομέρειε πώς αυτή η αλληλεγγύη θα λάβει σάρκα και οστά. Πώς θα παραμείνει απλώς γράμμα και περιεχομένου. Για την αλληλεγγύη νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Έχουμε το γραφείο του για το άσυλο, θα το, έχουμε στήσει, θα το στήσουμε σε λίγο. Ε, πολλά χρήματα για το Frontex και τον έλεγχο των συνόρων. Ε, αυξήθηκαν τα χρήματα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε το πρόγραμμα αυτό με τις εννέα χώρες που αναφέρατε ε, και ελπίζω να εμπλακούν και περισσότερες χώρες, αλλά είναι μια καλή αρχή. Και θα δούμε πώς θα το μονιμοποιήσουμε, αν θέλετε, αυτό το πρόγραμμα, ε, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Θα κάνω και προτάσεις για το πώς θα ενδυναμώσουμε τη Frontex ε, ως ονούπο και θα πιέσουμε τις, κράτες, ε, χώρες μέλη να συμμετάσχουν και να, να, υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια του πακέτου ασύλου και μετανάστευση Όλες οι χώρες έχουν δεσμευτεί, αλλά ξέρετε κι εσείς κι εγώ ότι οι τάσεις έτσι, στις διάφορες χώρες διαφέρουν. Ε, διαφέρει και η θέλησή τους να προχωρήσουν. θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα και με συγκεκριμένο τρόπο να τους δείξουμε την αλληλεγγύη. Η Κομισιόν θα υλοποιήσει αυτά τα εργαλεία σε μεγάλο αριθμό. Ευχαριστώ κύριε Μωράς. Κύριε Μάνστρομ, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, η αλληλεγγύη είναι από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να σας απασχολήσουν. Αλλά στην ε, εισαγωγή σας μιλήσατε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς ε, θα είστε τώρα η πρώτη επίτροπος όπου μοιράζεται το χαρτοφυλάκιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά ε, έχετε το Eurodac, τους αρατές σώματος, τα δεδομένα των ε, επιβατών και μια σειρά άλλων θεμάτων που περιλαμβάνουν εκτός από την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς πώ θα ασχοληθείτε με την ουσία των προβλημάτων αυτών βεβαίως θα είστε σε επαφή με τον συνάδελφό σα, αλλά αυτό νομίζω θα είναι μια μόνιμη πηγή συγκρούσεων ενδεχομένως. Παράδειγμα, Eurodac για τα δακτυλικά αποτυπώματα, για να σας πω πώς, λειτουργεί. Ε, θα υπάρχει μια βάση δεδομένων με δακτυλικά αποτυπώματα για τη μετανάστευση και θα έχουν πρόσβαση εκεί διοκτικέ αρχές. Πώς θα το λύσετε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά ε, πάντα χωρίς να λησμονείτε και την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Μωρέ. Ναι, είναι ένας νέος πράγματι επιμερισμός του χαρτοφυλακίου το αποφάσισε ο κύριος Παρόσο ίσως για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκόλμη. χρειάζεται τόσο πολλή δουλειά ε, ότι, ε, που θα χρειαστούν δύο γυναίκες για να την κάνουν ε, ή και τρεις άντρες και είπε η κυρία Ρέντινγκ ότι θα συνεργαστεί μαζί μας έτσι ώστε ε, όλες οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι υπό το πρίσμα των ε, θεμελιδών δικαιωμάτων και προσβλέπω σε πολύ σερή συνεργασία. Ποια είναι η διαφορά τώρα. Έχουμε τη ε, Λισαβόνα και συναπόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που πολλές από τις αποφάσεις που θα ενταχθούν στη Λισαβόνα θα σα διαβιβαστούν και θα είναι αντικείμενο συναπόφασης. Ξέρω πόσο ε, ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο και πόσο προσιλωμένοι είσαστε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίω μπορεί να προκύψουν συγκρούσει, το είπατε κι εσεί, αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα το χειριστούμε και για όσου με γνωρίζετε. Ξέρετε ότι όλη μου την πολιτική ζωή την έχω αφιερώσει στα ανθρώπινα δικαιώματα και πάντα ε, θέλω να αφήνω το στίγμα μου ε, και σε αυτό το χαρτοφυλάκιο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματική ερώτηση του κ. Μωράης. Ακόμα και για δύο γυναίκες θα είναι πολλές οι προκλήσεις. Μία από αυτές θα βρίσκεται στον πυρήνα των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσετε. Πρόκειται για την... Πρόκειται αυτό που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από ε, Γάλλο Υπουργό να λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR. Υπάρχει το πρόβλημα της ε, επεξεργασίας των PNR των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσείς Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα. Η κυρία Μάλμστρομ. Ναι, το PNR είναι ένα, είναι ένα παράδειγμα. Η η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, μια συμφωνία για τα PNR και ε, σύντομα θα γίνει αξιολόγηση του κόστους, του όφελους ε, των διαστάσεων προστασίας των δεδομένων. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλες αυτές τις πτυχές πρωτού προχωρήσουμε πιο πέρα. Και δεσμεύομαι να κάνω μια επισκόπηση των δομών που έχουμε εντό ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε τι έχουμε, τι λείπει, τι περιτεύει, πώς μπορούμε να τα οργανώσουμε αυτά με καλύτερο τρόπο. Και η αναλογικότητα, η αποτελεσματικότητα ε, ε, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Πλάσετ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ σήμερα. Το σύστημα ασύλου θα πρέπει να δημιουργηθεί χωρίς καθυστέρηση, λέτε. Ε, η ερώτησή μου είναι, στα πλαίσια της ε, καλύτερης νομοθεσίας μπορείτε να μου αναφέρετε μία οδηγία που θα πρέπει να αποτελέσει την ε, βάση του πακέτου ασύλου. Ε, δεύτερη ερώτηση. Εννοείται ότι ε, αυξάνεται συνεχώς η πίεση της λαθρομετανάστευσης. Η πιο αυστηρή έλεγχη στα σύνορα δεν μπορεί να είναι ο, ε, ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις ροές. Εσείς τι πρωτοβουλίες θα υιοθετήσετε σχετικά με την λαθρομετανάστευση και όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, η πρόσβαση σε καλό εργατικό δυναμικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2005 ε, ανακοινώθηκαν ε, σχετικά μέτρα. Η Κομισιόν όμω δεν έχει, υιοθετήσει ακόμα σχετική, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα σχετική οδηγία. Θα υιοθετήσετε τέτοια οδηγία στα πλαίσια αυτά. Ε, πολλές ερωτήσεις για δύο λεπτά. Πρώτη ερώτηση είναι, νομίζω ότι πράγματι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει ένα συνολικό πακέτο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί. Ε, αλλά φυσικά η ε, οι συνθήκες υποδοχής ε, θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι, θα πρέπει να είναι ίσες ε, και προβλέψιμες οι συνθήκες υποδοχής. Θα πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη να μπορούν να ανταποκριθούν ε, στα μέτρα αυτά. Έχουμε πολλά διαφορετικά στήματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε κοινό, κοινή πολιτική ασύλου θα πρέπει να, οι συνθήκες υποδοχής να είναι οι ίδιες και αυτό αποτελεί κομμάτι των πολιτικών αυτών. Η μετανάστευση είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Από τον καιρό του Αδάμ και της Εύας ε, γίνεται μετανάστευση. Αν θέλουμε όμω πολιτική μετανάστε... ασύλου που να είναι ε, αξιόπιστη, όπω είπα στον κύριο Μπαζούτη, θα πρέπει να ελέγξουμε και τα σύνορά μα. Ε, και χρειαζόμαστε διάφορα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. Ήδη σα ανέφερα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν τα επαναλάβω γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Θα πρέπει όμω να διασφαλίσουμε τι νόμιμε οδού προ την Ευρώπη. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε ρυθμιστούν και θα πρέπει να είναι ε, αξιόπιστε και να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνία των κρατών μελών. Θα προτείνω λοιπόν διάφορε οδηγίε. Μία θα ε, αφορά του εποχιακού εργάτε ε, και επίσης ε, μια οδηγία που να διευκολύνει τις ε, μεγάλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, που θα στέλνουν προσωπικό στην Ευρώπη. Αυτές τις προτάσεις θα τις υποβάλω πολύ σύντομα, τώρα στις αρχές της χρονιάς δηλαδή, για να τις συζητήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ανέφερα τους πιο αυστηρούς ελέγχους ε, συνόρων που δεν μπορούν να αποτελέσουν τη μόνη λύση αλλά είναι πολύ σημαντική. Είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε το ρόλο της ε, Frontex και καλά κάνετε. Η, αυτή τη στιγμή η Frontex ε, δεν έχει δικό της εξοπλισμό και τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση να την υποστηρίξουν. Έχετε σκοπό να παρουσιάσετε ένα υποχρεωτικό σύστημα για τη συμμετοχή των κρατών μελών ε, στη Frontex ή ε, προτείνετε η Frontex να έχει δικό της εξοπλισμό. Ε, αν όχι, γιατί όχι και αν ναι, πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Πώς βλέπετε την αφοσίωση αυτή τη στιγμή των κρατών μελών προς τη Frontex. Μιλήσατε για αλληλεγγύη. Πώς προτείνετε να ε, αυξήσετε την ε, πολιτική βούληση των κρατών μελών ε, να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, ήδη τώρα στις αρχές του χρόνου με την εμφύλαξη της έγκρισής σας θα υποβάλω πρόταση για την μεταρρύθμιση της Frontex που θα περιλαμβάνει πρόταση για ειδικευμένα τμήματα. Θα αναφέρει πώς η Frontex θα μπορεί στο μέλλον να συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες και θα προτείνω η Frontex να μπορεί να αγοράζει το δικό της εξοπλισμό, να προμηθεύει το δικό της εξοπλισμό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις της. Ε, αυτό θα την διευκολύνει διότι συχνά τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις αλλά τελικά κάνουν πίσω και έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να οργανώσουμε τέτοιες επιχειρήσεις. Η Frontex θα πρέπει να έχει εργατικό δυναμικό, ε, τεχνογνωσία για να ε, ε, για να μπορεί να συμμετέχει στον έλεγχο των συνόρων. την αλληλεγγύη την συζητήσαμε με τον κύριο Μπιζούτιλ. Έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας. Έχουμε οικονομικά, πολιτικά, θα έχουμε, το γραφείο ασύλου, έχουμε το πρόγραμμα τη Μάλτα και θα εργαστώ για να γίνει αυτό ένα πιο σταθερό κομμάτι ε, του όλου πλαισίου και θα πρέπει να συνεργαστούμε για να δούμε πώς θα περάσουν αυτά από το Συμβούλιο. Ξέρω τι δυσκολίε, αλλά είναι και η μόνη οδός που γνωρίζω που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σαρχεντίνη, ευχαριστώ πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Μάστρομ, η ομάδα των Πρασίνων έχει να αποθέσει πολύ μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες στο πρόσωπό σας για τη μετανάστευση και το άσυλο. Έχουμε όμως και μία ερώτηση. Στο παρελθόν δυστυχώς ζήσαμε προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση, την νόμιμη μετανάστευση, να ε, έχουν οδηγηθεί σε εμπλοκή στο Συμβούλιο. Εσείς τι φρονείτε γι' αυτό και γενικότερα πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα της εμπλοκής στο Συμβούλιο ε, προτάσεων, ε, αν σας τύχει, ε, για νόμιμη μετανάστευση. Και μετά το πρόγραμμα της πολιτικής το 2005 για την νόμιμη μετανάστευση δεν είδαμε πολλά χειροπιαστά αποτελέσματα. Και αναφέρομαι εδώ στη οδηγία για την ενιαία αδειοδότηση μάλλον άδεια παραμονής εποχιακών εργαζομένων έχετε συγκεκριμένα σχέδια για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη και σας ευχαριστώ για την ε, εμπιστοσύνη σας. Δεν είμαι υπεράνθρωπη, θα κάνω ό,τι μπορώ. Στο πρόγραμμα Στοκχόλ είναι σαφές και μάλιστα την εποχή του Άμστερνταμ ήταν σαφές ότι τα κράτη-μέλη θέλουν ε, και δεσμεύονται να δημιουργήσουν προγράμματα και για την νόμιμη μετανάστευση. Ε, θέλουμε ανθρώπου στην Ευρώπη. Έχουμε οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή βέβαια, αλλά θα περάσει. Και χρειαζόμαστε ήδη σε διάφορου τομεί, και φυσικά όχι με τον ίδιο βαθμό σε όλε τι χώρε, χρειαζόμαστε όμω ανθρώπου. Ε, αυτό είναι σαφέ. Και στη στρατηγική Ευρώπη για το 2020 θα υπάρχει αυτό το θέμα. Ε, πρέπει να έχουμε λοιπόν νόμιμους τρόπους για να έρθει κανείς στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένας τρόπος επίσης για να καταπολεμήσει και την λαθρομετανάστευση. Να αφήσουμε ε, την νόμιμη μετανάστευση να προχωρήσει για την ενία άδεια παραμονή. Ε, είχε κολλήσει εδώ και καιρό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχουν οι συνθήκε και να ξέρει ο κόσμο, αν έρθει νόμιμα στην Ευρώπη, έχει μια δέσμη δικαιωμάτων. Ε, και η οποία είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό για να προσελκύσουμε ανθρώπου στην Ευρώπη. Θα είναι επωφελέ για την οικονομία μα. υπάρχει επιχειρηματικότητα χάρη σε αυτό. Θα εμπλουτιστούν οι χώρε μα πολιτιστικά επίση με τι εμπειρίε των ανθρώπων αυτών. Νομίζω, όπω σα είπα, ότι υπάρχουν τρει προτάσει, ε, θα ξεκινήσουμε με τους εποχικούς ε, εργαζόμενους και επίση ε, την οδηγία για τι εταιρείε και θα υπάρξει και μια άλλη οδηγία για τους μαθητευόμενους. Στο Συμβούλιο θα προχωρήσουμε αυτά τα πακέτα και θα συνεργαστούμε και μαζί σα για να τα υλοποιήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό, όπω είπα, για την Ευρώπη και την οικονομία τη. Είναι σημαντικό για την ενίσχυση και την ανάπτυξη άλλων χωρών να έχουμε συμφωνίε με τρίτε χώρε. Αν θέλουν αν θέλουμε να μα βοηθήσουν για να καταπολεμήσουμε την λαθρομετανάστευση, θα πρέπει να του δώσουμε και δυνατότητα να έρχονται νόμιμα. Και βεβαίω θα αξιολογήσουμε και την πλέον κάρτα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι σε λειτουργία. Αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα. Θα ασχοληθώ λοιπόν με αυτό το θέμα το πρώτο εξάμεινο. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Θα δώσω τώρα το δικαίωμά μου, αν θέλετε, στην κυρία Φλότχα. Η δεύτερη, λοιπόν, η δευτερολογία θα γίνει από την κυρία Φλότχα. Ευχαριστώ για τους ε, νόμιμους μετανάστες στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι συχνά πέφτουν θύματα ε, διακρίσεων, ε, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Έρχομαι από την Καλαβρία ε, με άλλους συναδέλφους και οι εργάτες που δουλεύουν στη Γεωργία ε, δεν έχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα εκεί. Εσείς είπατε ότι θέλετε να αφήσετε το στίγμα σας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ ξέρω ότι έχετε να κάνετε πάρα πολλά. Την περασμένη ε, εβδομάδα ήρθε εδώ πέρα ο διευθυντής της Frontex. Θέλετε να ενδυναμώσετε τη Frontex, να εμπλέξετε τα κράτη-μέλη στη δουλειά της Frontex, ε, αλλά αν μιλήσατε ε, με τον διευθυντή, ε, θα σας πει ότι είναι λες και η Frontex θέλει απλώς να διώξει εμπορεύματα. Για... Αντιμετωπίσει τους ανθρώπους σαν εμπορεύματα. Ε, μιλάω τώρα για τους μετανάστες που είτε είναι ετούνται σε άσυλο ή όχι. Θα πρέπει να υποφελούνται εν πάση περιπτώσει από τα δικαιώματά τους. Πώς θα το εξασφαλίσετε αυτό ούτως ώστε να τα καταφέρετε. Κυρία Μάλστρομ, πώς θα λειτουργήσετε. Γνωρίζω το πρόβλημα, λέει η υποψήφια επίτροπο. όταν λέτε για όταν μιλάτε για τα δικαιώματα των ελεύθερων μεταναστών ή των νόμιων μεταναστών, φυσικά θα πρέπει να υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Όλων των ανθρώπων. Για την ε, άδεια των εποχικών εργαζομένων. Ε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην συναδελφό σας. Η Ευρώπη, η Ιταλία και άλλοι χώρες θα πρέπει να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα ε, γιατί υπάρχουν θύματα διακίνησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, οι διακινητέ αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν εμπορεύματα. Δεν τους αφήνουν ούτε δικαιώματα, ούτε δεν τους δίνουν μισθό. Πέφτουν και θύματα, α πούμε, έτσι ταραχών ε, και εξεγέρσεων στις τοπικέ κοινωνίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, υπερασπίζοντας τα σύνορα, να σεβαστεί την αρχή της μη επαναπρόθεσης, τα ατομικά δικαιώματα των ετούν τον άσυλο και να εξασφαλίσει ότι κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να κάνει αίτηση για άσυλο. Και φυσικά, εν συνεχεία, η διαδικασία και η απάντηση το ναι ή το όχι είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η Ευρώπη έχει αυτό την υποχρέωση και θα εξασφαλίσω μαζί με την κυρία Ρέντινγκ ότι η Frontex και όλες οι άλλες υπηρεσίες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπίζονται αυτά τα δικαιώματα είναι καθήκον μας. Ο κύριος Κίρκοπ. Πρόεδρε, ε, κύριε Πέτροπε, τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε κάποια γεγονότα ε, για τα θέματα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας να κυριαρχούν. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης τονίζει ότι χρειάζεται συνολική και διευρωπαϊκή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου, του διεθνούς, ε, στον κύπερνο χώρο, τη διακίνηση ανθρώπων και γενικά χρειάζεται ισχυρότερη καταπολέμηση και της διαφοράς. Τα κράτη-μέλη έχουν υποδομή, έχουν δίκτυα, έχουν οργανισμούς και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, προτίθεστε στο μέλλον να προχωρήσετε στον τομέα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και εδώ και διεθνώς με τους φίλους μας για να βεβαιωθούμε ότι όσο τα κάνουμε αυτά ε, έχετε πάντα στο μυαλό σας την έννοια της αναλογικότητας στην απάντηση που δίνει η Ευρώπη σε αυτά τα θέματα. Η κυρία Μάνστρο. Ευχαριστώ κυρία Μάλιστα, μάλιστα αυτή είναι μια από τις προτεραιότητες με την οποία θα ασχοληθώ πολύ σύντομα. Η εσωτερική στρατηγική ασφάλεια την χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τι απειλέ τρομοκρατία, οργανωμένου εγκλήματο και τι άλλε που αναφέρατε. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια πράγματα. Θα πρέπει όμω να αξιολογήσουμε πιο ολοκληρωμένα τα μέσα που έχουμε για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Και θέλω μια συνολική επισκόπηση των μέσων που έχουμε κατά τη τρομοκρατία όταν μιλάμε για την ε, συνεργασία μας με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, ε, την νομοθεσία, τις πολιτικές, ε, τα ταμεία, για να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μπορεί κάτι να μας λείπει, μπορεί να υπάρχει επικάλυψη εργασιών που θα πρέπει να εξαλειφθεί. Την αξιολόγηση αυτή θα την υποβάλω στην Επιτροπή σας πολύ σύντομα. Όσον αφορά τα νέα συστήματα πληροφορικής. Πάντα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την αρχή τη αναλογικότητα, το κόστος, την προστιθέμενη αξία που επιφέρουν και με το σεβασμό της ε, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και όπως σας είπα, θα εξετάσω ακριβώς με αυτά τα γυαλιά, με αυτό το φακό ε, τα μέσα αυτά. Και όσον αφορά την τρομοκρατία, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα μέσα που έχουμε για να έχουμε καλή πρόληψη, προστασία και ανταπόκριση. Έχουμε διάφορα νομοθετικά μέτρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τα θύματα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα στον τομέα αυτό, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με τα θύματα της τρομοκρατίας. Αυτό θα προταθεί στα πλαίσια της εσωτερικής ε, στρατηγικής ε, ασφαλείας. Ο κύριος Κάκο πάλι. Ναι, με ναι, καθησυχάστε με την απάντηση αυτή, άσχετα όμως με το πόσες ε, γυναίκες, ε, ε, όσες γυναίκες όμως και να ασχολούνται στο τομέα αυτό, η Επίτροπος ως δυνατή γυναίκα μπορεί να με καθησυχάσει ότι η ίδια αναλογικότητα που αναφέραμε πριν λίγο θα ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της νομοθεσίας που θα επιβληθεί στα κράτη-μέλη στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης του εγκλήματος και ότι θα συνεχίζει να υπάρχει στο επίκεντρο η αυξημένη συνεργασία λαμβάνοντα υπόψη τι εθνικέ προτεραιότητε ε, και ενδεχόμενε εξαιρέσει. Ε, και συμφωνείτε μαζί μου ότι μία γενική ενιαία ε, πολιτική μπορεί να μην είναι πάντα αποτελεσματική ή πρακτική. Όπως είπατε, στον τομέα της τρομοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολλά νομοθετικά μέσα. Η επιχειρησιακή ευθύνη ανήκει στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί μόνο να συντονίζει και να βλέπει πώς μπορεί να ενισχύσει ε, τα μέτρα και έχουμε κάνει πολλά στον τομέα αυτόν. Όταν μιλάω λοιπόν για μια γενική επισκόπηση, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να υποβάλω νέε νομοθετικέ προτάσεις, σημαίνει ότι θέλω να έχω μια επισκόπηση που θα είναι χρήσιμη με τον προκάτοχο μου τον κύριο Μπαρό έχει συζητήσει το θέμα αυτό η Επιτροπή σας. Ε, τα μέσα που έχουμε, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με πιο έξυπνο τρόπο, μήπως μπορούμε να ε, ε, ξεφορτωθούμε κάποια περιτά πράγματα, μήπως υπάρχουν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να συλληρωθούν. Αυτό είμαι διατημένη να το συζητήσω μαζί σας τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Σταφάρης eh, Ευχαριστώ κύριε Μάλστρομ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε για τα θέματα ασύλου. Δεν θέλω γενικές διακήρυξεις, αλλά συγκεκριμένες δηλώσεις. Ο διευθυντής της Frontex ήρθε την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο και μας μίλησε για συμφωνίες με τη Λιβύη και μας είπε ότι είναι και ευπρόσδεκτη είδηση. Αλλά εσπρέσω λίγο καιρό μετά επιβεβαίωσε αυτά που εμείς ήδη υποπτευόμαστε, τη μεταχείριση δηλαδή επιφυλάσσει η Λιβύη στους ε, ανθρώπους αυτούς, τους παρατάει στη Σαχάρα περίπου στη μοίρα τους και μέχρι θάνατο αντιμετωπίζουν. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά, θα αναθεωρήσετε την εντολή του Frontex για να επανέλθουμε σε μια παλαιά ανθρωπιστική παράδοση που είναι η διάσωση στο πέλαγος για παράδειγμα. Πώς θα... Ε, προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην επαναπροωθείται κανείς ε, σε χώρες που δεν σέβονται τη ε, συνθήκη της Γενέβης για τις πρόσφυγες και διώκεται με βάση την προέλευσή του, το φίλο, τη φιλή κτλ. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω εάν κατάλαβα ακριβώς την ερώτησή σας, αλλά θα επανέλθετε στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη της ε, όπως και όλοι οι πολίτες ε, και οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Εγώ θα ενισχύσω με τη Frontex, θα πρέπει να ξαναδώ και το δίκαιο της θαλάσσης, γιατί είναι δύσκολο για τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για τους ορισμούς. Ε, κυκλοφορούν κάποιες προτάσεις στο Συμβούλιο και θα σταλούν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα καθήκοντα των κρατών μελών και της Frontex όταν δρούν ε, ε, στη θάλασσα. Πραγματικά αυτό θα βοηθήσει. Η αρχή της μη επανοπρόθεσης είναι διεθνή σύμβαση και εμεί ως δημοκρατικά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευόμεθα και είμαστε υποχρεωμένοι να διαβεβαιώσουμε ότι θα προστατεύουμε εκείνους που ε, διώκονται από καταστολή και υφίστανται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποφέρουν σε δικτατορικά καθεστώτα και φεύγουν για να ξεφύγουν για να σώσουν τη ζωή τους. Για τη Μεσόγειο όμως είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς αν είναι οικονομική μετανάστευση ή όχι. Όπως πολλοί Ευρωπαίοι πριν από έναν αιώνα που έψαχναν μια καλύτερη ζωή γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη ένδια και φτώχεια. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας μου πριν από 100 χρόνια έφυγε από τη ε, Σουηδία γιατί ήταν τόσο φτωχοί και πήγαν στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, ζητώντας καλύτερη μοίρα και βοήθησαν να οικοδομηθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, για να κάνουν την τύχη τους. Για το θέμα της Λιβύης. Και βέβαια ε, θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τη Λιβύη, να συζητούμε. Είναι σημαντική η χώρα γείτον. Ε, είναι χώρα διέλευση και στέλνει και κόσμο και δεν είναι εύκολο γιατί είναι ακριβώ ο ορισμό της δημοκρατικής χώρας η Λιβύη. Θα πρέπει να βρούμε όμω έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Ξέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε μια προσέγγιση και από την προηγούμενη Προεδρία προ τη Λιβύη ε, με πάρα πάρα πολύ μικρά και αργά βήματα αλλά θα πρέπει να συνεργαζόμαστε επαναλαμβάνω με τους ε, Λιβύους και να δούμε πώ θα ενισχύσουμε πάντα τη δέσμευση που έχουμε και εμείς και εκείνοι να σέβονται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνεργάζονται με την ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες που είναι παρούσα στη Λιβύη ε, για να δούμε τι γίνεται σε έκτακτες περιστάσεις. Εύκολα δεν είναι όλα αυτά, θα είναι μακράς πνοής και μικρά βήματα, πάντως θα πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Ξανά ο κύριος Ταβάρες. Κυρία Μάλστρομ. Μιλήσαμε για προβλήματα. Ας μιλήσουμε τώρα για λύσεις. Μία από τις αποτελεσματικές λύσεις για τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο είναι η επανεγκατάστασή τους. Κάτι που είναι διαφορετικό ε, από τη μεταφορά των μεταναστών από ευρωπαϊκή χώρα σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτούς τους επιτρέπουμε να έρθουν στην επικράτειά μας από τις χώρες. Ο Υπουργό Μετανάστευση τη Σουηδία λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να υποδεχθεί 100.000 ε, πρόσφυγε. Αυτή τη στιγμή ε, εγκαθιστούμε 5.000 το χρόνο. Πώ μπορούμε να φτάσουμε στι 100.000. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ. σω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δημιουργήσει ε, μια νέα δομή που θα ασχολούνταν αποκλειστικά με αυτό. Με επανεγκατάσταση των προσφύγων. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα. Έπειτα, τα δικαιώματα των νομίμων μεταναστών που θα, θα πρέπει να μοιάζουν ε, με των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουν και δικαίωμα ψήφου. Για πέστε μας κυρία Μάλστρομ. Ίσως να μην κατάλαβα καλά την ερώτησή σας γιατί ήταν, ε, άγγιξε πάρα πολλά ερωτήματα. Ε, είσαστε εισηγητή για την οδηγία επανεγκατάσταση, κύριε Ταβάρε, και περιμένω τι απόψει σα. Γιατί η επανεγκατάσταση είναι μία από τις πολλές λύσεις. Πολλές χώρες έχουν ήδη εμπλακεί, κάποιες άλλες μπορούν να κάνουν περισσότερα. Ε, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες της, έτσι. Ε, και κάποιες άλλες τρίτες χώρες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Είναι ένα τμήμα τη ευρύτερη λύση για επανεκατάσταση, ούτω ώστε να δώσουμε καταφύγιο σε αυτού του ανθρώπου και να ε, αναλάβουμε κι εμεί ω Ευρώπη τι ευθύνε μα. Ευχαριστώ. Ο κ. Μποργκέτσιο Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, εκτίμησα πάρα πολύ την ε, ορθολογική και μη ιδεολογική προσέγγισή σας. Έτσι βλέπετε τη μελλοντική σας δραστηριότητα και τα θέματα μετανάστευσης. Παρ' όλα αυτά δεν κατάλαβα πολύ καλά. Και αν θέλετε εξηγήστε μου το λίγο περισσότερο. Δεν κατάλαβα τι θα γίνει με αυτή την οδηγία για τις πολυεθνικές. Δεν το πιάσα αυτό. Συχνά στην Επιτροπή μας ακούμε τους εκπροσώπους χωρών ε, της Βόρειας Ευρώπης, όπως η δική σας χώρα, που στυλιτεύουν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανθρωπιστική μεταχείριση, ε, ειδικά σε θέματα ασύλου. Αυτές οι ίδιες χώρες όμως είναι εντελώς απούσες όταν έρχεται η ώρα για να μοιραστούμε την προσπάθεια ε, για χώρες που κάνουν χώρες όπως η δική μου, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ισπανία. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα μόνες μας, μόνες αυτές οι χώρες. Προβλήματα υποδοχής ε, μεταναστών, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την επίπτωση της παρουσίας των μεταναστών στις χώρες μας και των ετούντων άσυλο. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο, η Επίτροπος ε, Φεραίρο Βάλνερ ε, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ε, από τον Πρόεδρο δεν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν και 27 χώρες με συγκεκριμένο τρόπο και αυτό σημαίνει και στα έξοδα. Γιατί αυτό είναι το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε στο διατάφτα, πώς μοιραζόμαστε και το βάρος, το οικονομικό. Κυρία Μάλστρομ. Η Ευρωπαϊκή, Η Ευρωπαϊκή Ένωση Όμω, ε, συχνά συγχαίρει τον εαυτό της ε, για το ότι είναι ο βασικό φορέα που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον κόσμο. Γι' αυτό ε, έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από δικτατορικά καθεστώτα κτλ. Και συμφωνώ μαζί σα ότι κάποιε χώρε αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και άλλες λιγότερη. Αλλά πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη γίνει. Έχουμε μιλήσει για το μοίρασμα των ευθυνών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη πίεση σε κάποιες χώρες της Μεσογείου, αλλά και οι περισσότεροι ε, πρόσφυγες έρχονται αεροπορικά, έρχονται και, με άλλους τρόπους, δεν έρχονται μόνο μέσω της Μεσογείου. Ξέρω ότι η Μεσόγειος βρίσκεται υποπίεση και ε, ανέφερα κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, με τη Frontex, με προγράμματα επανεκατάσταση ε, με τρόπους συνεργασίας με τρίτες ε, χώρες ε, στην περιοχή της Μεσογείου. Θέλω να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, θέλω όμως να τονίσουμε, θέλω να τονίσω όμως ότι έχουμε και διεθνή υποχρέωση να δεχτούμε τους ανθρώπους ε, που ζητούν άσυλο και να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους. Ε, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Μπάτιν για την συμπληρωματική ερώτηση, όχι. Ο κύριος Πορκέσιο. Ελπίζω λοιπόν αυτή τη φορά να απαντήσετε στη συγκεκριμένη μου ερώτηση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει τα δικαιώματα στο πλαίσιο του ασύλου και τα ανθρωπιστικά δικαιώματα ε, κατά την επανεγκατάσταση. Αλλά σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να επιμεριστούν οι προσπάθειες και στους 27. Και γιατί τελικά το ανθρωπιστικό βάρος ε, και το οικονομικό βάρος πέφτει σε τρεις-τέσσερις χώρες. Η Frontex μας ανακοίνωσε, και αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον για όλους, μία αναδιοργάνωση εσωτερική της. υπάρχουν πολλά πράγματα που έθιξαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ θα σας πω δύο μόνο. Πρώτον, υπάρχει ένα πολύ λεπτό θέμα της του επαναπατρισμού που το διαχειρίζεται, που το έχει αναλάβει η Frontex και το χρηματοδοτούν όλες ε, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των επιμέρους κρατών μελών. Ε, το πρόβλημα όμως είναι ότι στην πραγματικότητα βαραίνει περισσότερες, κάποιες λίγες χώρες όπως τη δική μου. Έπειτα, τα κέντρα ε, υποδοχής θα πρέπει, ε, πιστεύετε, να τα διαχειρίζεται η Frontex. Κυρία Μάλστρομ, ευχαριστώ κύριε Μποργέζιο. Πιστεύω ότι η Frontex και στην πρόταση που θα κάνω, που δεν έχω κάνει ακόμα όμως, γιατί πρέπει να την ετοιμάσω, θα προτείνω λοιπόν ότι η Frontex θα αγοράσει τον εξοπλισμό της για να είναι καλύτερα εξοπλισμένη ε, για τις κοινέ επιχειρήσεις. Η τελική ευθύνη όμως για τα σύνορα είναι ευθύνη των κρατών μελών. Η Frontex μπορεί να συντονίσει και να βοηθήσει. Η Frontex μπορεί να βοηθήσει και τα κράτη-μέλη για τον, ε, για τον ε, επαναπατρισμό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει σωστή εξέταση αν το συγκεκριμένο άτομο, άτομο δεν θέλει να κάνει αίτηση ασύλου, αν η διαδικασία έχει γίνει σωστά και μπορεί να σταλεί πίσω χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, χωρίς να υποστεί κακομεταχείριση. Με βάση την αρχή τη μη επαναπρόθεση. Η Frontex εκεί μπορεί να βοηθήσει. Αλλά την τελική ευθύνη πάντα την έχουν τα κράτη-μέλη. Ποιο είναι επόμενο, η κυρία Μόρβαε. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομες ερωτήσεις έχω δύο, παρακαλώ να μου απαντήσετε. Στις 23 Οκτωβρίου του 2006 στη Βουδαπέστη υπήρξε μία διαδήλωση με μεγάλες ε, παραβιάσεις. Ε, η διαδήλωση αυτή ε, κατεστάλλει βία με πολλούς τραυματίες. Το είδαν και οι τουρίστες και είχαμε και μαρτυρίες τουριστών στη Βουδαπέστη τότε που υπήρξαν και τις συνέπειες. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να ρωτήσω. Στη συνέχεια ακολούθησαν ε, διώξεις. Ε, η αστυνομία έκανε διάφορες έρευνες, έψαχνε σε σπίτια με γυναίκες μόνες τους, ώρες ολόκληρες χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς πληροφορίες. Γενικά, ο πρόεδρος διακόπτη, κυρία Μόρπαϊ. Ναι, εσείς τι θα κάνετε για να μην επαναληφθεί τέτοια κατάσταση ξανά. Ευχαριστώ κυρία Μορβέ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Ενθυμούμε τα γεγονότα του 2006 και γνωρίζω επίσης ότι κάποιος Σουηδός υπουργό ήταν παρόν τότε και έζησε τη γεγονότα αυτά τη βία. Κάτι λέει η κυρία Μορβά εκτός μικροφώνου, δυστυχώς δεν ακούγεται. Αλλά βεβαίως αυτό είναι θέμα των Ουγγρικών αρχών να διερευνήσουν αν έκανε κατάχρηση εξουσίας, υπέρβαση καθήκοντος η αστυνομία ή αν έδρασε με τρόπο αντίθετο προς την Ουγγρική νομοθεσία. Και το άλλο που αναφέρατε είναι εθνικό ζήτημα. Δεν μπορεί να το σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Και πάλι κυρία Μορβάη. Bonds, then I, I guess I... Όχι. Ο κύριος Μποντς. Κυρία Μάλμστρομ, δεν με καθεσίγασα αυτά που μας λέτε. Το αντίθετο μάλιστα, έχω θορυβηθεί βαθύτατα. Γιατί και εσείς μιλάτε υπέρ της μαζικής ε, μετανάστευσης με διάφορα ε, επιχειρήματα τύπου γύρανσης και ανταγωνισμού. Έχει ολόκληρα εκατομμύρια μιλιούνια ανέργους η Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνουν δουλειά και δεν βρίσκουν και εσείς έρχεστε εδώ και πρεσβεύετε μαζική μετανάστευση και τη δικαιολογείτε κιόλας. Τα προβλήματα τα ξέρετε στις μεγαλοπόλεις, ε, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, το Λονδίνο, στο Μάλμεο, στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ, στις μεγάλες πόλεις. Τεράστια προβλήματα με τη μαζική μετανάστευση. Και έρχεστε εδώ και μας ε, λέτε ε, νέα κύματα μετανάστευσης. Όταν σας ακούω τέτοια πράγματα ανησυχώ τόσο πολύ. Ελπίζω να μην αναλάβετε επίτροπος εσωτερικών ε, υποθέσεων. Γιατί αν σας βάλουν σε αυτή τη θέση θα γεμίσουμε ε, και άλλους μετανάστες και δεν επιτρέπεται τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ. Εξαρτάται από χώρα σε χώρα. Αλλά όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε ε, στο μέλλον θα χρειαστούν εργάτε. Εξαρτάται, ανάμεσα στις, ε, εξαρτάται από το μέσα τομέα και από τι ανάγκε τη κάθε χώρα. Χώρας. Αλλά για να διατηρήσουμε τι οικονομίε μα και για να πληρώσουμε τα, τη συντάξη των ηλικιωμένων και να εξασφαλίσουμε το σύστημα ευημερία, χρειαζόμαστε την νόμιμη μετανάστευση. Ε, μετανάστευση. Φυσικά δεν είναι η μόνη λύση ε, στα οικονομικά προβλήματα που έχουμε. Είναι τμήμα της λύσης όμως. Και έχουν γίνει πάρα πολλές στατιστικές, ε, δημογραφικές και έρευνες που το δείχνουν αυτό. Φυσικά θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιου τομεί θα δεχτούμε αυτούς τους μετανάστες. Η κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίσει. Αλλά ως Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει μια επισκόπηση, θα κάνουμε μια επισκόπηση. Έπειτα, οι άνθρωποι αυτοί το, για το πώς θα ενταχθούν στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, αυτό είναι βασικά θέμα των κρατών μελών ε, να το εξασφαλίσουν. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση, λοιπόν θα έχετε ένα χαρτοφυλάκιο και ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου σας θα είναι να βάλετε τάξη στην πολιτική μετανάστευση στην Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, Ηράκλειο έργο. Ε, ξέρω τις δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη, ε, τις σημερινές δημογραφικές τάσεις. Ε, με βάση αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θαύματα σε αυτόν τον τομέα. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, ε, κυρία Μάλστρομ, ότι σε κάποιο βαθμό χρειαζόμαστε μετανάστες στην Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό. Στην εισαγωγική σας δήλωση είπατε ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια κατάσταση όπου όλοι θα κερδίσουν. Φυσικά αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξή. Τι ιδέες, τι σχέδια έχετε για την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα είναι τελικά σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Γιατί θα γίνει τελικά πόλεμος για τους μισθούς. Θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, και αυτοί θα κερδίσουν από τη μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πάουερ. Πολύ επίκαιρη ερώτησή σας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν όλοι. Κάποιοι από αυτού που έρχονται θα επιστρέψουν στις χώρες τους, θα έχουμε κυκλική μετανάστευση, άλλοι θα θέλουν να μείνουν. Αυτό θα το αποφασίζει το κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να λαμβάνονται υπόψη και κάποιες ηθικές πτυχές. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαφυγής εγκεφάλων, brain drain. Θα συνεργαστώ με τον συνάδελφο που θα είναι υπεύθυνο για την απασχόληση για να φροντίσουμε αυτοί που έρχονται, είτε έρχονται βραχυπρόθεσμα είτε μόνιμα, να έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα στην αγορά εργασίας με δίκαιους μισθούς, σε δίκαιες συνθήκες, χωρίς να ανταγωνίζονται αθέμητα τους άλλους. Έχουμε ε, διάφορες οδηγίες που ρυθμίζουν το θέμα αυτό. Θα πρέπει να ληφθεί λοιπόν υπόψη και είναι κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο στενή συνεργασίας για να μην πετύχουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Δευτερολογία η κυρία Πόσκουρτ. Μπάουερ πάλι. Η κυρία Μπάουερ πάλι. Θα επανέλθω και αργότερα. Ε, μία συμπληρωματική ερώτηση έχουμε κάποιον κανονισμό που αφορά τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε εργοδότες που απασχολούν λάθρομετανάστες. Πώς ε, μπορείτε να εφαρμόσετε την νομική ευθύνη των υπεργολάβων. Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία, δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να την εφαρμόσουν ήδη τώρα και αυτό αποτελεί κομμάτι της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης. Να έχουμε νόμιμη μετανάστευση, αλλά να ελέγχουμε και την εμπορία ανθρώπων, διότι Πολύ συχνά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων φτάνουν στην Ευρώπη με πολλές υποσχέσεις και ζουν υπό απαράδεκτες συνθήκες. Βλέπουμε τις συνέπειες στην Ιταλία και αλλού. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν οι εργοδότες να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για σωστή απασχόληση. Θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία στις εθνικές αρχές, θα πρέπει να είναι ένα εθνικό σύστημα. Οι εργοδότες, εάν παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς, ε, σημαίνει ότι παραβαίνουν τον νόμο, ε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο τα κράτη-μέρη να εφαρμόσουν ήδη τώρα την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Καλημέρα σας, κυρία Μάνστον. Πολλές γυναίκες προσπαθούν να διαφύγουν από διώξεις που έχουν να κάνουν με το φίλο τους, όπως είναι ο ακροτηριασμός των γεννητικών τους οργάνων ή η κατανακαστική ε, γάμη. Αλλά δεν τους δίνουν άσυλο, διότι δεν διέπονται τα θέματα αυτά από το άσυλο, με εξαίρεση τη δική σας χώρα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις αρχές του 2010 το γραφείο του ασύλου θα ιδρυθεί και θα κατασταθεί στη Μάλτα και χρειάζεται και τους απαραίτητους πόρους. Μπορείτε να μας αναφέρετε τρία συγκεκριμένα μέτρα ε, που ε, θα είναι τομείς δράσης του Γραφείου Ασύλου για προστασία των γυναικών που ε, διώκονται και γι' αυτό φεύγουν από τις χώρες τους γιατί παραβιάζονται τα ειδικά ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Μάστρο. Thank you for Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Γνωρίζουμε ότι παγκοσμίω ε, οι περισσότεροι μετανάστες είναι γυναίκες. Όχι μόνο στην Ευρώπη, η πλειονότητα των μεταναστών είναι γυναίκες. και θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη ευαισθησία ως και προς το φύλλο και στην πολιτική ασύλου και μετανάστευση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα για ευάλωτες ομάδες, ε, γυναίκες, παιδιά, έγκυες γυναίκες, ε, ανθρώπους με αναπηρία κτλ. Ωστόσο, το Γραφείο Ασύλου και οι γενικές πολιτικές θα χρειαστεί να αναλύσουν αυτή τη διάσταση του φύλου. Δηλαδή πώς μπορούμε κατά την υποδοχή να έχουμε ειδική μέρημνα για γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση, ε, να έχουν μια ειδική προσοχή ε, για αποκατάσταση της υγείας τους, ε, άνδρες και γυναίκες ενδεχομένως να διαμένουν χωριστά, οι γυναίκες με παιδιά να έχουν ειδική αντιμετώπιση και φροντίδα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και πώς επίσης πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη. Εν πάση ε, θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο ε, της εντολής του Γραφείου Ασύλου, αλλά και της γενικής εντολής μας όταν νομοθετούμε για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, διότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί σε όλους τους τομείς νομοθεσίας. Και συνεργαζόμαστε ήδη προς την κατεύθυνση αυτή με την κυρία Ρέντινγκ και για το ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όντως θα πρέπει οι γυναίκες αυτές να προστατεύονται στην Ευρώπη και λαμβάνουμε ήδη μέτρα για να καταπολεμήσουμε ε, αυτή την κατάσταση και στο μέλλον οπωσδήποτε. Η κυρία Μποσκούρτ. Uh, female genital ο ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ένα πρόβλημα αντινόμενο στην Ευρώπη, έχει οξυνθεί ακριβώς γιατί έχουμε ε, πολλέ μετανάστριες από χώρε που υπάρχουν τέτοιες πρακτικές. Ε, εάν το κάνουμε αυτό προτεραιότητα και προσπαθήσουμε να εκριζώσουμε αυτή την κατάσταση θα στείλουμε και ένα σαφέ μήνυμα ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η πρακτική παγκοσμίω. Τι ρόλο θα διαδραματίσετε εσεί σε αυτό τον κλάδο, πώ βλέπετε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση ακριβώς του αγροτηρισμού των ε, γεννητικών οργάνων στις γυναίκες. Απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ξεκάθαρη ε, νομική εξουσία για θέματα ενδοοικογενειακής βίας ή τέτοιων φαινομένων που εκεί μπορούν να ενταχθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έχει αρχίσει να ετοιμάζει μία ανακοίνωση για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και γνωρίζω ότι είναι και προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο, υπάρχουν και άλλες τρομερές ε, βιαιότητε ε, που ε, υφίστανται οι γυναίκε στην Ευρώπη, ενδοοικογενειακή βία. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο προληπτικά να εργαστούμε. Υπάρχουν ήδη πολύ καλά παραδείγματα από το πρόγραμμα Δάφνη που συνεργαζόμαστε με τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, θρησκευτικού ηγέτες για να σταματήσουν την πρακτική αυτή ορισμένες εθνωτικές ομάδες και, και ορισμένες οικογένειες που προέρχονται ε, από συγκεκριμένες χώρες. Πραγματικά είναι τρομερά αυτά που υφίστανται τα δεινά ε, γυναίκες και τα κορίτσια και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακολίνο. Ναι, εδώ, εδώ είμαι. Μιλήσατε στην αρχική σας παρουσίαση ε, την απέτηση να ε, ασχοληθούμε με τους διάφορους οργανισμούς agencies. Υπάρχει και ο οργανισμός της Λισαβόνας για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι ένα πρόβλημα που οξύνεται όλο και περισσότερο. Οι νέοι καταναλώνουν και περισσότερο ψυχότροπες ουσίες ε, και σε συνδυασμό με ενόπνευμα είναι ανεπανόρθωτες οι ζημίες που προκαλούνται. Στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρόσφατα ασχολήθηκε στο πρόγραμμα της Στοχόλμης και με την καταπολέμηση και με την πρόληψη από αυτού. Εσείς τι θα κάνετε, ε, πώς θα καθοδηγήσετε το παρατηρητήριο προς την κατεύθυνση αυτή και πώς προτίθεστε να συνεργαστείτε με την κυρία Ρέντινγκ για μια τέτοια συμφωνία, αλλά και με τον Επίτροπο για την προστασία του καταναλωτή, για να προστατεύουμε πραγματικά τους Ευρωπαίους πολίτες. Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα που θίγεται κύριε Τσακολίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι έχει κάνει αρκετά. Τα κράτη-μέλη φυσικά έχουν την τελική ευθύνη και έχουμε διαφορετική νομοθεσία. Έχουμε προχωρήσει λίγο στο θέμα του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά. Έχουμε την υπηρεσία για τα ναρκωτικά και τον εθισμό και έχουμε και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πολύ ευχαρίστω να συνεργαστώ μαζί σας για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βρούμε μέτρα για να συντονίσουμε τη δουλειά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όπως είπατε είναι ένα θέμα που άπτεται πτυχών υγεία, ε, εγκληματικότητας, οργανωμένου εγκλήματος, ε, διακίνησης ναρκωτικών πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινότητες, ε, την κοινωνία, ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα αυτό. Γνωρίζω καλά το πρόγραμμα, το πρόβλημα αυτό. Δεν βλέπω όμως ε, τα, να έχει τα μέσα αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το αντιμετωπίσει. Ε, θα το συστήσω όμως και με τους άλλους αρμόδιους επιτρόπους, ε, τον κύριο Ντόλ και την κυρία Ρέντινγκ, όπως είπατε. Ε, μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος αυτού και μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι θα πρέπει να εργαστούμε κυρίως σε τοπικό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Τζακολίνο. Κάτι που συνδέεται με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι ο υπερπληθυσμός των φυλακών. Σε πολλές ε, χώρες μέλη το 1 τρίτο των φυλακισμένων ε, είναι ξένοι και το 1 τρίτο έχει προβλήματα αλκοόλ, ναρκωτικών, σοβαρότατα προβλήματα που επιβάλλουν την παροχή ε, εξειδικευμένη ιατρικής ε, φροντίδας. Το πρόγραμμα της Ε, πώς ε, παρεμβαίνει θα διευρύνουμε, θα φτιάξουμε νέες φυλακέ, θα διευρύνουμε τις υπάρχουσες. Πώς θα εξασφαλίσουμε την κοινωνική ένταξη, ούτω ώστε να δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία σε ανθρώπους ε, που πέρασαν από τη φυλακή και πώς θα τους εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ζωή. Τι προγράμματα θα υλοποιήσετε μετά από τις διατάξεις που περιλαμβάνει αυτό το έγγραφο που ονομάζεται το κείμενο της Στοκχόλμης. Το πρόγραμμα, συγγνώμη, της Στοκχόλμης. Κύριε Ιακολίνο, ε, ομολογώ ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ότι θα πρέπει να το προσέξουμε όλο ιδιαίτερω. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε, μπορούμε να δώσουμε κάποια εργαλεία, ε, θα πρέπει να δώσουμε και κάποια χρηματοδότηση σε συγκεκριμένα προγράμματα, να ανταλλάξουμε ιδέε, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα που αναφέρατε αντιμετωπίζονται καλύτερα εθνικά ή τοπικά, στι τοπικέ κοινωνίε. Και με βάση την αρχή τη αναλογικότητα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη αντιμετώπιση ε, ενδεχομένως σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Ε, βεβαίως θα πρέπει ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανταλλάξουμε εμπειρίε. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε συγκεκριμένα νομοθετικά εργαλεία ή απτά εργαλεία που μπορούμε να προτείνουμε για αυτό το θέμα, παρότι ε, ομολογώ ότι όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο κύριος Κρίστιανσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν και εργάζονται παράνομα στην Ευρώπη. Πολλοί ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μια καλύτερη ζωή και ορισμένοι ξεγελάστηκαν ότι θα ζήσουν ε, μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Ε, παραμένουν παράνομα στην Ευρώπη και εφόσον παραμένουν παράνομα δεν έχουν ε, δικαίωμα ασφάλισης, δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, δεν πληρώνουν φόρους κτλ. Με τον τρόπο που ε, δουλεύουν και εργάζονται και παραμένουν εδώ είναι μοντέρνοι σκλάβοι και επομένως ε, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ε, υπάρχει όμως και μια τεράστια ζήτηση για λαθρομετανάστες. θα κάνετε για να μειωθεί αυτή η ζήτηση για λαθρομετανάστες. Σας ευχαριστώ με συγκινεί πραγματικά πολύ ο τρόπος ε, που με κοιτάτε και που περιμένετε από μένα να επιλύσω αυτά τα τεράστια προβλήματα. Η εμπιστοσύνη που μου έχετε με συγκινεί. Ε, η Κομισιόν και η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει. Έχει... Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ορισμένοι έρχονται στην Ευρώπη ε, γιατί τους ξεγέλασαν ότι θα βρουν θαυμάσιες δουλειές και ορισμένοι ζουν σε άθλιες συνθήκε σε, σε απαράδεκτους οίκους ανοχής ε, ως ε, μοντέρνοι σεξουαλικοί σκλάβοι. Θα πρέπει να βρούμε ε, τα νομικά εργαλεία για τους εποχιακού εργαζόμενους, για τι εταιρείε ανάλογα με τι ανάγκες των κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε νομοθεσία, ούτως ώστε αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη τελικά να έρχονται νόμιμα και να έχουν αυτά τα δικαιώματα τα οποία είναι ισοδύναμα με αυτά των Ευρωπαίων πολιτών. Και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις όμορες χώρες, ούτω ώστε να εμπλακούν και αυτές. Ε, να τους ενημερώνουν, να τους δίνουν και άλλα μέσα, να υπάρχουν α, ε, συμφωνίες ε, κινητικότητας με τις χώρες αυτές για να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή έρθουν σε μια χώρα, τα νόμιμα δικαιώματα που έχουν ε, ε, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ε, στη δική μου χώρα και στη δική σας χώρα γίνεται μια έντονη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να δώσουμε πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι, θα, ότι προβλέπεται να υπάρξει κοινή νομοθεσία στην Ευρώπη για αυτούς τους ξένους υπηκόους. Ο κύριος Κρίστιανσεν. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε για, τις, ε, για την ε, οδηγία για τις κυρώσεις που ε, προσπαθεί να τιμωρήσει τον εργοδότη και όχι τον εργαζόμενο. Εσείς πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι εργοδότες στο μέλλον δεν μπορούν να προσλαμβάνουν τέτοιους παράνομους εργαζομένους και να μένουν ατιμόρυτοι και πώς θα εφαρμόσουμε σωστά ως Ευρώπη αυτή την οδηγία. Αυτό θα πρέπει να γίνει, λέει η κυρία Μάλστρομ, Α, κυρία Μάστομα, πρέπει να πω το όνομά σα, ότι είναι η σειρά σα, λέει να απαντήσετε. Ε, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που γίνεται πάντα. Η, η, η, η Κομισιόν πάντα εποπτεύει την ε, εφαρμογή μιας οδηγίας. Δεν θα πρέπει στην Ευρώπη ε, οι εργοδότες να χρησιμοποιούν του διακινητέ ω εργαλεία. Θα πρέπει να γίνει ένα έλεγχο εθνικά καταρχάς ε, με βάση τα συστήματα των κρατών μελών, άλλη κομισιόν. Είναι ο θεματοφύλακα των συνθηκών και θα πρέπει να ελέγξει ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τι οδηγίε που αποφασίσαμε. Θα γίνει με τον τρόπο δηλαδή που, γίνεται πάντα για τι οδηγίε και θα διστάσω να παραπέμψω τα κράτη-μέλη στο δικαστήριο σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση αυτή τη οδη... ή άλλων οδηγιών. Thank you. Mrs. Σίπελ. Ευχαριστώ, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλμστρομ, θα ήθελα να σας κάνω μια γενική ερώτηση αρχής και ακούγοντας την εισαγωγή σας νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε πολύ σύντομα. Μπορείτε να δεσμευτείτε τυπικά και επίσημα ότι σε συνεργασία με την κυρία Ρέντινγκ και το Συμβούλιο θα έρχεστε τακτικά στην Επιτροπή μας για να συζητούμε θέματα διεθνών συμφωνιών. Ε, με τρόπο ε, πλήρη, ε, άμεσο και αμέσως να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 218 της Συνθήκης Λισαβόνας. Και δύο λόγια για το SWIFT. Ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχετε υπόψη σας για την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα του SWIFT ως μέτρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και ένα τελευταίο, αν έχουμε χρόνο ακόμα, από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα τρία σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για σας για το SWIFT ή κατά την άποψή σας πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν. Ναι, τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Ναι, δεσμεύομαι εάν ε, οριστώ να ε, έρχομαι στην Επιτροπή σας όπως έκανε και ο προκατοχός μου. Με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας ούτως ή άλλως θα έχουμε πολλά θέματα που απαιτούν συναπόφαση. Θα εμφανίζομαι λοιπόν συχνά στην Επιτροπή σας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό. Πρόκειται για υπόσχεση. Όσον αφορά το SWIFT, έχουμε μια προσωρινή εννιάμινη συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα μου έχουν δοθεί κάποια σαφή παραδείγματα της χρησιμότητας του SWIFT. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο στον εντοπισμό χρηματοδότησης για τρομοκράτες. Ε, ε, πριν ε, λίγο καιρό υπήρξε αποστολή προς τη Washington όπου συζητήθηκε το θέμα αυτό και θα ήθελα οι αρχέ επιβολή του νόμου να σα δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα προσπαθήσω να τα βρω αυτά για να δείτε τη χρησιμότητα. Έχω κάποια ε, παραδείγματα. Κάποια άτομα καταδικάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο ε, Σεπτέμβριο κάτι που και επίσης επέτρεψε το σύστημα SWIFT τις ε, γερμανικές αρχές να προλάβουν μια επίθεση το 2007 και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν προλάβει πολλές ε, επιθέσεις ε, με τον εντοπισμό των ε, χρηματοδοτικών ροών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το μέλλον του SWIFT, θα συζητηθεί αυτό και θα επανέλθουμε με νέες πληροφορίες ιδιαίτερα ε, αυτά που αφορούν μια πιο μόνιμη συμφωνία SWIFT. Αυτό θα πρέπει να ε, συμφωνηθεί μαζί με το Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ η προστασία των δεδομένων και αν μπορούμε να βελτιώσουμε την προσωρινή συμφωνία ε, ακόμα περισσότερο στον τομέα αυτό, αυτό θα είναι θετικό. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Θα ήθελα να διευρύνω το ερωτηματολόγιο. Αναφέρατε πριν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει στρατηγική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ευρωπαϊκή στρατηγική κάθε φορά μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις ε, λαμβάνονται κάποια μεμονωμένα μέτρα. Μετά τις ε, επιθέσεις του Σεπτεμβρίου του 2001 και μετά την ε, τρομοκρατική επίθεση τώρα πριν τα Χριστούγεννα αναφέρεται συνέχεια το θέμα, το θέμα αυτό. Οι εμπειρογνώμονες όμως αφισβητούν τα θέματα αυτά και έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τα τεχνικά μέτρα η απάντηση στο πρόβλημα. Γι' αυτό ρωτώ ήδη πριν το αναφέρατε αυτό, ε, ποιοι θα πρέπει να είναι οι βασικοί πυλώνες μια ενιαίας στρατηγική για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και τι μέτρα δεν έχουν εισαχθεί ακόμα και θα πρέπει να εξεταστούν πιο προσεκτικά. Η κυρία Μάλμστρομ, κυρία Σίπελ. Ίσως να υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη μετάφραση. Εγώ τόνισα τουλάχιστον μία φορά ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από την κατακαιρματισμένη αυτή προσέγγιση της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θέλω μία επισκόπηση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αυτό αφορά και την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, τις διάφορες πολιτικές, τα διάφορα ταμεία, τις διάφορες οδηγίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά και θα το κάνω αυτό σε συνεργασία με την κυρία Ρέντινγκ. Θα εξετάσω την όλη αρχιτεκτονική ανταλλαγή πληροφοριών και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια γενική επισκόπηση, να δούμε εάν λείπει κάτι, εάν υπάρχει κάτι περιττό ε, θα ε, αξιολογήσουμε λοιπόν ε, τα μέτρα. Το θέμα είναι η αποτελεσματικότητα, το κόστος και η προστιθέμενη αξία που θα επιφέρουν τα μέτρα αυτά. Εντός της στρατηγικής, στα πλαίσια της στρατηγικής ασφαλείας θα σας υποβάλω συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια, τις καλύτερες ευχές μου και καλή σας τύχη. Θα ήθελα να επανέλθω στο Frontex περισσότερες λεπτομέρειες για να καταλάβουμε. Ο Frontex είναι ένας οργανισμός κυρίως συντονισμού, ανάλυσης, επαναπροώθησης και ε, εκπαίδευσης της ακτοφυλακής. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υποκατάστατο εθνικών αρχών. Ποτέ. Άρα τι θέλουμε να κάνουμε εμείς με το Frontex. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, κυρία μου, είναι να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες που έχει και να φροντίσουμε όταν είναι πολύ κρίσιμες οι καταστάσεις ε, να υπάρχει μια δυνατότητα και ε, ε, ένας κατάλογος προθέσεων, καλών προθέσεων ή ε, συγκεκριμένη συνεισφορά σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υλικό, υποδομή, τι θα πρέπει ο καθένας να δίνει στο Frontex. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Όταν προβληματιζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή και πριν αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε το κανονισμό του 2007 του 2004. Τελειώνω, Πρόεδρε. θα συνεχίσω στη συνέχεια. Τι προτείνετε να κάνετε και το Κοινοβούλιο πώς θα συμμετέχει εκεί. Ευχαριστώ πολύ η απάντηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Frontex έχει κάνει ανάλυση και αξιολόγηση και έχει καταθέσει και μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί ο οργανισμός αυτός. Όπως είπατε είναι οργανισμός, agency, συντονιστικό ρόλο έχει και υποβοηθητικό, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη φύλαξη των συνόρων στο σύνολό της. Ε, πολλά βασίζονται στην αλληλεγγύη στα πλαίσια του Frontex. Είναι εύκολη στα λόγια η αλληλεγγύη, καμιά φορά είναι πιο δύσκολη στα έργα και συγκεκριμένες δράσεις. Εγώ θα κάνω ε, την πρόταση για ενίσχυση του Frontex όπως είπατε, θα ε, τους δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσουν τον εξοπλισμό τους οι ίδιοι για να μην εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη κατά περίπτωση ότι έχουν ευχαρίστηση. Ε, θα έχουν ειδική ε, κατεύθυνση θα συνεργάζονται με ε, τη ε, φύλαξη των συνόρων και τη Eurosur που ελπίζω να έρθει κατά τη διάρκεια της παρουσιτίας και θα συνεχίσουμε ακριβώς και την εκπαίδευση των ε, φυλάκων, των συνοριοφυλάκων, της ακτοφυλακής για την αρχή της και με το Γραφείο Σύλλου και βεβαίως θα συνεργάζονται και με τις τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες επανεισδοχής. Και θα φροντίσω να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Βεβαίω θα συνεργάζονται και με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ και την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία Ασύλου ε, για συντονισμό στι τρίτες χώρες όπως είναι η Λιβύη. Ορίστε λοιπόν ε, συγκεκριμένα μέτρα για να προχωρήσουμε. Αλλά εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ίδια τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και στις επιχειρήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Αυτό εμείς δεν μπορούμε παρά να το διευκολύνουμε, να τους αναγκάσουμε, να τους διατάξουμε, δεν μπορούμε. Ευχαριστώ κύριος Δίας Δεμέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Frontex εργάζεται ήδη και συνεργάζεται με το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση και την ύπατη αρμοσία. Έχει 83 εκατομμύρια ευρώ και 222 υπαλλήλους και με πολύ μεγάλη δυσκολία εκτελούν τον προϋπολογισμό. Πολύ μεγάλη. Αυτό που θέλει είναι να ε, αλλάξει προς ανατολισμό και να κοιτάει προς τον νότο. Γιατί είδαμε τραγωδίες στην Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Ιταλία, στην Ισπανία. Στο νότο είναι το πρόβλημα. Και υπάρχει λοιπόν εδώ μια ανισότητα. Ε, κυρία Επίτροπε, ε, υποψήφια, λέτε θέλετε να αγοράσει εξοπλισμό. Τι να αγοράσει. Ε, αυτό που χρειάζεται μόνο είναι συστήματα διαβιβάσεων τηλεπικοινωνιακά για να υπάρχει συμβατότητα. 2007-2013 τι θα τους πούμε, πάρτε αεροπλάνα, καράβια, ελικόπτερα, να το κάνει τι η Frontex. Ένα μικρό κρατος μέλος δεν έχει τόσο εξοπλισμό. Ε, κυρία Μάλστρομ, ναι είναι πρόβλημα αυτό. Το, η Frontex έχει λεφτά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί υπάρχει αβεβαιότητα. Αν θα λάβουν χώρα οι επιχειρήσεις, αν θα συμμετάσχουν ή όχι τα κράτη-μέλη, αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Ε, η Frontex θα μπορούσε λοιπόν να αγοράσει εξοπλισμό και μηχανήματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αναλύσουμε εάν είναι υποφελή σε σχέση με το κόστος τους ούτως ώστε να γίνει πιο ανεξάρτητη από τα κράτη-μέλη τα οποία κατοδοκούν συμμετέχουν ή όχι στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα λυθούν υπόψη σε λίγους μήνες ή λίγες εβδομάδες όταν παρουσιάσω την πρότασή μου για την ενίσχυση της Frontex. Κυρία Μπάουερ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε με μεγάλη τιμή θα επανέλθω για δεύτερη φορά και θα εκπροσωπήσω την ε, Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών εκ μέρους του ΕΛΚ. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της διακίνησης ατόμων. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα και του προγράμματος Στοκχόλμης. Και εκ μέρους της ε, Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Ξέρω ότι το 80% των θυμάτων ε, της διακίνησης είναι γυναίκες ή νεαρά κορίτσια. Και παρά τις ευρωπαϊκές μας προσπάθειες, παρόλα αυτά αυξάνεται η διακίνηση ατόμων ε, και ο αριθμός των θυμάτων επίσης αυξάνεται. Επομένως, τι νομικά εργαλεία θα θέλετε να δημιουργήσετε, κυρία μου, για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει να συμφωνήσει βεβαίω και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εσεί τι σκοπεύετε να κάνετε για να προστατεύσετε τα θύματα, για να μην πέσουν θύματα μια δεύτερη φορά αυτέ οι γυναίκε. Ποιε είναι οι προθέσει σα, ποια είναι τα σχέδιά σα και πώς μπορεί να μειωθεί η ζήτηση για τις γυναίκες αυτές, για τα κορίτσια αυτά. Κυρία Μάλστρομ, ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία ε, με συγκινούν και προσωπικά πολύ έντονα. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα φρικαλαίο έγκλημα και οι περισσότερες γυναίκες, ε, τα κορίτσια και τα, παιδι και τα αγόρια ακόμα, είναι θύματα. Δεν μπορώ να φανταστώ μια μεγαλύτερη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από το να τα πουλάμε ως σεξουαλικούς σκλάβους. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν εξίσου σοβαρά και να αντιμετωπίσουν αυτό το, αυτή την τάση ως ε, έγκλημα με αντίστοιχες κυρώσεις. Υπάρχει στο Συμβούλιο μια πρόοδος, μέχρι στιγμής δεν έχουμε συμφωνήσει, αλλά παρόλα θα έχουμε προχωρήσει. Θα ε, θα κάνω τώρα μία πρόταση έτσι, πιο σύμφωνη με το πνεύμα της Λισαβόνας για τη διακίνηση, αλλά και την σεξουαλική ε, εκμετάλλευση των παιδιών. Και ελπίζω με τη συναπόφαση που τώρα έχουμε και την στεναρή δέσμευση του Κοινοβουλίου και, σε, και πολλών κρατών μελών, να το πούμε και αυτό, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για αυτή την οδηγία, γιατί πραγματικά είναι αφρικόδε έγκλημα. Επίση, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα θύματα και την ε, αποκατάσταση των θυμάτων. Αυτό είναι ένα βήμα μετά. Ε, μπλέκονται εδώ και πολλοί άλλοι. Ε, και αυτό σχετίζεται με, με μέτρα που θα πρέπει να προωθηθούν, αλλά που δεν τα έχω εγώ απόλυτα στη διάθεσή μου με βάση το χαρτοφυλακιό μου. Ε, γιατί έχουν μια εξωτερική διάσταση αυτά τα ζητήματα και μια διάσταση ε, πολιτικής, ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με μη κυβερνητικού οργανισμού. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά καλά προγράμματα στη Μολδαβία, α πούμε, για την αποκατάσταση αυτών των νέων γυναικών και προσπαθούμε να του δώσουμε μια δουλειά και να τι βοηθήσουμε να ενταχθούν στι κοινωνίε. Ευχαριστώ. Ξανά κύριε Μπάουερ. Ευχαριστώ. Μου αρέσει αυτή η δέσμευση που δείχνετε για αυτό το τομέα. Θα μπορούσα να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Αν λάβουμε υπόψη την εμπειρία μας ε, σε αυτόν τον τομέα. Ξέρουμε ότι πολλέ ε, γενικές διευθύνσει εξετάζουν αυτό το θέμα, αλλά προς το παρόν δεν έχει υπάρξει συντονισμό. Τι θα γίνει με τους εθνικούς συντονιστέ. Ε, ο καθένας δρά στον τομέα του, αλλά δεν, δρά, δεν δρούνε με έναν ευρωπαϊκά συντονισμένο τρόπο. Θέλετε να υπάρξει ένας ευρωπαίος συντονιστή για αυτό το θέμα. Είσαστε υπέρ μια τέτοια ιδέα. Η κυρία Μάλστρομ. Ναι, είναι η απάντηση. Φυσικά, λέει η κυρία Μάλστρομ. Και ελπίζω ότι ο Ευρωπαίος ε, συντονιστής αυτός να εντάσσεται, να υπάγεται σε μένα και να συνεργάζεται με τους εθνικούς συντονιστές. Και το πρόγραμμα Στοκχόλμης και η μελλοντική πολιτική επιστροφής θα βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε κυρία Μπάουερ. Θα πρέπει να συντονίσουμε τα εργαλεία μας και τις πολιτικές μας και αυτό θα κάνουμε με αυτές τις οδηγίες ε, και την ε, εσωτερική στρατηγική ασφάλειας. Θα συνεργαστούμε με τις άλλες γενικές διευθύνσεις, γιατί πολύ σωστά ε, το ίδιο πρόβλημα εξετάζεται και από άλλες γενικές διευθύνσεις από, άλλο πρίσμα. Παραδείγματος χάρη η Lady άστον, είναι και αυτή στην αρμόδια. Κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, το θέμα μου αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ούτω ώστε κάθε τμήμα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση να υλοποιηθεί. Επίση, σε τι θα δώσετε προτεραιότητα, σε τι μέτρο θα δώσουν προτεραιότητα οι υπηρεσίε σα και τι προτεραιότητα θα δώσετε στην επιστροφή των ε, λάθρο μεταναστών στις χώρες τους. Ευχαριστώ. Κυρία Μάλστρομ, το σύμφωνο για τη μετανάστευση θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να αξιολογηθεί του χρόνου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα που είναι ήδη λειτουργικά, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί όλα. Θα πρέπει να, εγώ να καθορίσω κάποιες προτεραιότητες, καταρχάς για το άσυλο. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πακέτο ασύλου. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στο... και θα είναι δύσκολα στο Συμβούλιο. Δεν είμαι αφελής, το ξέρω. Αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε κοινού κανόνες για τους ετούντες άσυλο. Ε, και για να βάλουμε και λίγη τάξη ε, στα εθνικά συστήματα, ούτω ώστε να αποφύγουμε τις ανθρώπινες τραγωδίες. Επίσης όμως κοστίζει να αφήνουμε τον κόσμο ε, να περιμένει πάρα πολύ πριν υποβάλει την αίτηση. Τώρα για τη λαθρομετανάστευση. Έχω αναφέρει ήδη κάποιες προτεραιότητες. Θα πρέπει να προσφέρουμε νόμιμα εργαλεία για αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Θα ενδυναμώσω τη Frontex, όπως εξήγησα στους συναδέλφους σας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες. Νομίζω το νέο γραφείο ε, για το άσυλο στη Βαλέτα που θα είναι λειτουργικό από φέτος το φθινόπωρο θα είναι και αυτό χρήσιμο για να βοηθήσει τις ε, τρίτες χώρες και να μας βοηθήσει για να μοιραστούμε, να μοιράσουμε τις ευθύνες μεταξύ των χωρών. Θα συνεχίσω και τη συζήτηση με τις τρίτες χώρες, κυρίως με τη Λιβύη και την Τουρκία, αλλά και με άλλες χώρες στην περιοχή, για να δούμε πώς μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες επανεισδοχής που οι οποίες συμφωνίες μας βοηθάνε να ελέγξουμε και την λαθρομετανάστευση. Η κυρία Ματιού μια δεύτερη φορά για αυτό το θέμα μιλήσατε, Φερρυπίν, για τη Λιβύη και για την Τουρκία. Μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι κάθε συμφωνία η οποία θα υπογραφεί με μια τρίτη χώρα θα περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο αποκλειστικά για τη μετανάστευση. Προφανώς. Με τις ενδιαφέρομενες χώρες, ε, με τη Λιβύη εμπροκειμένα και την Τουρκία, σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ε, είναι δύσκολες συζητήσεις, ειδικά με τη Λιβύη. Η η διαδικασία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα έχει ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι, χάρη στον κύριο Μπαρόζο, ο οποίο ε, ήθελε να πάει τον Νοέμβριο τον κύριο Μπαρό που ήθελε να πάει τον Νοέμβριο δεν μπόρεσε όμω. Ε, το θέμα είναι να δούμε πώ μπορούμε να συζητήσουμε με τι αρχέ τη Λιβύη. Αλλά το έχουμε στη μέση διάταξη αυτό το θέμα. Ε, φυσικά εξαρτάται από την κάστοτε κατάσταση τη τρίτη χώρα. Αλλά βέβαια θα το κάνουμε αυτό. Κυρία Η κυρία Ρέντινγκ θα έχει το βασικό ρόλο για την, ε, τα θέματα καταπολέμησης της, ε, των διακρίσεων. Πολλοί μετανάστες έχουν κάποια μορφή ε, αναπηρίας και επομένως ε, υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, όχι μόνο επειδή είναι μετανάστες, αλλά και επειδή έχουν αναπηρία. Νομίζω ότι όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να συνεργαστούν Εσεί πώς θα συνεργαστείτε με τη Vivian Redding και με την Επίτροπο Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, ούτω ώστε οι μετανάστε οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί ε, διακρίσει δεν θα πέσουν περαιτέρω θύματα λόγω τη ε, σεξουαλική του, σεξουαλικού του προσανατολισμού, ε, του φίλου του, τη ηλικία του, τη προέλευσή του. Ευχαριστώ, κυρία Λίν. ξέρω ότι σα ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα. φυσικά αυτό είναι κυρίως ευθύνη της ε, κυρίας Ρέντινγκ. Αλλά κάπως εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιό μου. Θα το συζητήσουμε. Είναι σαφές στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ότι οι ευάλωτες ομάδες, οι άνθρωποι με αναπηρίες, παιδιά, γυναίκες και άλλοι που υφίστανται ε, διακρίσεις και χρειάζονται περαιτέρω προστασία, θα εντοπιστούν ω ομάδες στις προτάσεις. Θα συνεργαστώ λοιπόν με την κυρία Ρέντιν και με άλλους επιτρόπους, ούτως ώστε αυτό το θέμα να ενταχθεί σε, ε, σε διάφορες προτάσεις που θα προωθήσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Λίν. Όπως γνωρίζετε, ήδη έχουμε σχέδιο πρότασης του Συμβουλίου. Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η ε, οδηγία κατά των διακρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αντιμετωπίζουν ε, διακρίσεις και μαζί με τους ε, συναδέλφους σας στην Επιτροπή θα ασκήσετε πίεση στο Συμβούλιο για να φροντίσετε την γρήγορη οριοθέτηση της οδηγίας αυτής. Ναι, κύριε Λίν, ε, στην προηγούμενη μου ιδιότητα Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για ε, Τη ε, ε, Σουηδική κυβέρνηση. Συνεργάστηκα πολύ στενά με τους συναδέρφους μου στη Σουηδική Προεδρία και ελπίζαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα. Δεν τα καταφέραμε τελικά. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητε. Ελπίζω ότι η Ισπανία το επόμενο τρίο προεδριών θα αναλάβει το θέμα διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί το θέμα. Θα συνεργαστώ στενά με την ε, Ισπανική Προεδρία και με το Συμβούλιο για να ε, περάσει η οδηγία αυτή και είναι σημαντική η οδηγία αυτή ε, όχι μόνο στα πλαίσια των εξωτερικών υποθέσεων αλλά στο, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Κιγιόμ. Θα επανέλθω κυρία μου στο θέμα της δέσμης του ασύλου. Στις γραπτές σας απαντήσεις είδα ότι είστε υπέρ μια ταχείας έγκρισης του θέματος αυτού, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει εμπλοκή για το Δουβλίνο 2, τον κανονισμό αυτό και για την υποδοχή των μεταναστών. Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη, και το είπατε, έχουν ε, εκφράσει οξύες επικρίσεις στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εναρμόνιση ε, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αρχίσει ακόμα να εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλετε να κάνετε για να σπάσει αυτή η εμπλοκή και να διατηρηθεί ο στόχος του 2012 για ένα κοινό καθεστώς ασύλου έτσι ώστε οι μετανάστες που διώκονται και διαφεύγουν να έχουν πρόσβαση ουσιαστική ε, στο άσυλο ε, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία κάνουν την αίτησή τους και να έχουν μια διεθνή προστασία. Ευχαριστώ κυρία Μάρσον. Ε, ναι κυρία Κιγιώμα, όπως λέτε είναι προτάσεις οι οποίες ε, είναι καθοδόν, αλλά όπως είπατε πάρα πολύ δύσκολο να εγκριθούν από το Συμβούλιο είναι συγκεκριμένες και γνωστές οι ευαισθησίες που υπάρχουν και προκαλούν δυσκολίες. Ωστόσο και το Συμβούλιο και όλα τα κρατημέλη συμφώνησαν για το πρόγραμμα της Στοχόλμης και το στόχο να ε, έχουμε μια κοινή ζώνη ασύλου το 2012 και οι πάντες έχουν υπογράψει αυτό το στόχο αυτό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχουν σωστές και αξιοπρεπείς συνθήκες και να επικρατούν οι ίδιες συνθήκες σε όλα τα κρατη δεν μπορώ παρά να χρησιμοποιήσω αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που μας δίνεται με την έγκριση του προγράμματος της Στοκχόλμης και τώρα ε, όλοι μπαίνουμε στο σύστημα της συναπόφασης και θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσετε και να εγκριθούν τελικά οι οδηγίες. Δεν σας κρύβω όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια αυτή και η συζήτηση που θα κάνουμε ε, από κοινού αν θέλουμε όμως να καταλήξουμε σε αυτό το στόχο, μια κοινή ζώνη το 2012, από τώρα πρέπει να αρχίσουμε και να επιταχύνουμε. Η κυρία Γκυγιόμ και πάλι. Αναμένοντας λοιπόν το 2012 και προς την ίδια κατεύθυνση ε, με τη δέσμευση που ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα η κυρία Ρέντινγκ που έχει φορτιστεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε εσείς να μας διαβεβαιώσετε ότι θα συνεχίσετε ε, να προσφέρετε στο δικαστήριο για ε, παραλήψεις και σε ε, περίπτωση επαναπροώθησης στη θάλασσα μεταναστών. Μιλώ λοιπόν για την προσφυγή επί παραλήψης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Μα και αυτό είναι ένα στοιχείο της δέσμης του πακέτου. Θα πρέπει ε, όλες οι χώρες να εφαρμόζουν εξίσου και με τον ίδιο τρόπο τις διατάξεις τις οποίες έχουν δεσμευτεί. Έχουν υπογράψει διεθνείς συμβάσεις, είναι συμβαλόμενα μέρη και θα πρέπει το δίκαιο να γίνεται σεβαστό και να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για διεθνή σύμφαση και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαχρυπνεί, αλλά και τα κράτη-μέλη να φροντίζουν να εφαρμόζονται όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κοέγιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε την Σεσίλια Μάλμστρομ, ξέρουμε ότι είναι ικανή και θέλουμε να αναφερθούμε στις προτεραιότητες. Η περιοχή Σέγγεν αποτελεί το κέντρο της ε, περιοχής ασφάλειας ε, ελευθερίας και είπατε ότι είναι σημαντικό να ελεγχθούν τα εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια εντός της Ευρώπης. Και έχουμε επίσης ε, το θέμα που θα έπρεπε να έχει ε, εφαρμοστεί το 2007. Έχουμε καθυστέρηση πάνω από 5 χρόνια και πάνω από 70.000 ευρώ έχουν διατεθεί πέρα από αυτά που έχουν διαθέσουν ε, τα κράτη-μέλη. Το ΣΥΣ αποτελεί προτεραιότητα για σας και πότε θα μπορέσει να εφαρμοστεί και εάν πάλι αποτύχουμε αυτό θα έχει συνέπειες. Η κυρία Μάλμστρεμ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέγιο. Το ΣΥΣ 2 είναι ένα θέμα που ανακάλυψα ότι θα κληρονομήσω με όλες τις δυσκολίες του. Ο εργολάβος δεν έχει πληρώσει τις ε, υποχρεώσεις του, δεν έχει ανταποκριθεί στα αναμενόμενα και δεν είναι ε, ιστορία με... δεν είναι μια ωραία ιστορία. Τέλος αυτής της εβδομάδας ε, και για κάποιες μέρες θα πρέπει ο εργολάβος να αποδείξει ότι ε, μπορεί να ολοκληρώσει το έργο και εάν ε, τα καταφέρουν ε, τότε θα συνεχίσουμε. Εάν όχι θα πρέπει να επανέλθω στο Συμβούλιο όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τους πω ότι όχι, λυπάμαι, δεν λειτουργεί η λύση αυτή. Θα πρέπει να εξετάσουμε την άλλακτική λύση. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα σε λίγες μέρες θα μπορέσουμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση κινούνται τα πράγματα διότι όπως είπατε, είναι σημαντικό για τη λειτουργία της ε, περιοχής Σέγγεν να λειτουργεί το ΣΥΣ 2. Πάντως αυτή η μακρά και ιστορία με τις πολλέ δυσκολίες ε, θα βρίσκεται στο γραφείο μου ε, τουλάχιστον ε, στην αρχή τη θητεία μου. Θα ενημερώνω το Κοινοβούλιο για το πώς προχωράμε. Εάν όλα πάνε καλά, στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον. Ο κύριος Κοέγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ΣΥΣ 2 είναι πράγματι μια δυσάρεστη περίπτωση, δεν είναι όμως η μόνη περίπτωση όπου έχουμε καθυστερήσεις και στο ΦΥΣ, έχουμε καθυστέρηση και στην πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη έχουμε καθυστερήσεις και θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Δεν έχει νόημα να ξεκινάμε, σε νέες περιπέ... να ξεκινάμε νέες περιπέτειες χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει τα προηγούμενα. Θα πρέπει λοιπόν, λοιπόν καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα προγράμματα που ε, έχουμε μαζί μας τα και χρόνια θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Ε, συμφωνείτε κυρία Μάλμστρομ. Ναι κύριε Κοέγιο και δεν έχω καν αναλάβει τα καθήκοντά μου ακόμα. Δεν μπορώ λοιπόν ε, να ε, αναφερθώ σε όλα όσα γίνονται. Ε, πάντως χρειαζόμαστε και το ΣΥΣ2, χρειαζόμαστε και το ΒΙΣ. Θα πρέπει όμως να έχουμε μία επισκόπηση των συστημάτων συλλογής πληροφοριών που έχουμε και που μπορεί να έχουμε στο μέλλον, ώστε να μην αναλαμβάνουμε βιαστικά την την πραγματοποίηση μεγάλων, ακριβών και πολύπλοκων συστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να περιμένουμε κάποιες ώρες, κάποιες μέρες να δούμε πώς θα πάει το ΣΥΣ2, διότι αποτελεί σημαντικό ε, θέμα. Νομίζουμε ότι έχει... Ε, ότι προχωράει πάλι, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά προτού να αρχίσουμε να συζητάμε άλλα πριν ξεκινήσουμε καινούργια προγράμματα θα πρέπει να λειτουργεί αυτό. σύμφωνο μαζί σα. Ευχαριστώ κύριο Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι Σεσίλια. Εδώ δεξιά σου. Γεια σου, καλημέρα, Καλώ όρισε, καλή σου τύχη. Μιλώ εξ ονόματο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και δύο πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει. Ε, πανέρχομαι στο θέμα του, της βίας του φίλου. Είπες ότι το θέμα της κοινοτικοποίησης αυτών των θεμάτων είναι περίπλοκο. Εσύ όμως θα μπορούσες συγκεκριμένα να σκεφτείς το άσυλο στα πλαίσια ακριβώς της ε, καταστολής και της βίας ε, αιτία το φίλο; ε, δηλαδή, εις βάρος των γυναικών. Για τις εξωτερικές σχέσεις τώρα θα πρότεινες εσύ μέτρα έτσι ώστε το στοιχείο του φίλου να συμπεριληφθεί στις συμφωνίες σύνδεσης. Και τέλος, πώς σκέφτεσαι να εργαστείς ε, με το παρατηρητήριο για την καταπολέμηση της ε, βίας κατά των γυναικών με το φύλλο και το Ινστιτούτο που εδρεύει στο Βίλνιους. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, πώς να το πω, ήδη έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τα μέτρα που ισχύουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ισχυθεί η συνεργασία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, αλλά αν χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία ε, και νομίζω ότι είναι προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας και του Τρίου. Ε, για τις άλλες ερωτήσεις σου θα προσπαθήσουμε σε όλα τα μέσα και όλα τα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, να εισάγουμε αυτό το στοιχείο του φύλου και να πούμε ότι έχουν ιδιαίτερη κατάσταση οι γυναίκες ε, που ζητούν άσυλο και είναι και πιο ευάλωτες και ενδεχομένω είναι θύματα βιασμού αλλά και κακοποιήσεων και βίας και ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων, όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Κατά τα άλλα, γνωρίζω και για τις άλλες συμφωνίες που δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό, είναι άλλων συναδέλφων, ε, θα προσπαθήσουν και εκείνοι να συμπεριλάβουν και το στοιχείο του φίλου στις αποφάσεις αυτές, ε, στις συμφωνίες με τις χώρες. Αυτό θα χρειαστεί να το παρακολουθεί και το Κοινοβούλιο και άλλοι και να φροντίζεται να εφαρμόζονται όλα αυτά. δουλειά υπάρχει, αλλά θα παρακαλέσω να ενισχυθεί η συνεργασία και θα φροντίσω κι εγώ να παρακολουθώ. Ε, ο κύριος Ρωμέβα, αυτό το τελευταίο που είπες, ποια είναι τα εργαλεία και τα μέσα, στα αγγλικά τώρα το παρατηρητήριο είναι από τα εργαλεία αυτά που σκέφτεσαι, γιατί ε, είναι υποστελεχωμένο και έχει πολύ περιορισμένο προπολογισμό. Δηλαδή χρειάζονται και περισσότερα πρόσωπα εκεί να εργάζονται και περισσότεροι πόροι. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις σχετικά με αυτό. Yes, I understand. Η κυρία Μάλσομ, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ε, δεν σας κατάλαβα καλά την πρώτη φορά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσω. Δεν ξέρω αρκετές λεπτομέρειες για να μπορέσω αυτή τη στιγμή να σας δώσω συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ όμως, θα πάρω τις πληροφορίες που μου δίνετε, θα εξετάσω το θέμα, θα επανέλθω αργότερα να δω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, διότι δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μάλμστρεμ, τονίσατε την πρόθεσή σας να αξιολογήσετε την παρούσα νομοθεσία για, την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της και να ασχοληθείτε με την Frontex, Europol και Cipol για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Αυτό μου φαίνεται πολύ λογικότερο από την μαζική συλλογή πληροφοριών. Είδαμε τι έγινε με τον Ομπάμα και την, ε, την, ε, την ε, τρομοκρατική επίθεση πριν τα Χριστούγεννα που έδειξε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η συλλογή των πληροφοριών. Την επισκόπηση αυτή θα την χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα συνεπές γενικό σχέδιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό και θα αποφύγετε το να κατακαιρματιστούν οι προσπάθειες. Έχουμε το ΣΥΣ, έχουμε το ΒΙΣ, ε, τα θέματα PNR, τα ε, στοιχεία εισόδου-εξόδου. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Η κυρία Μάλφστρομ, ναι, δύο παρατηρήσεις, ε, διότι είναι θέματα που θα συζητήσαμε νωρίτερα. Το σύνολο του προγράμματος της Στοκχόλμης και η εσωτερική στρατηγική ασφάλεια στο στόχο έχει να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. Άλλωστε είναι πολύ νέος ο τομέας αυτός ε, στην ε, ευρωπαϊκή συνεργασία. Ε, πρόσφατα γιορτάσαμε τη δεκαετία του. Ήταν λοιπόν κάπως κατακαιρματισμένες οι προσπάθειες. Χρειάζεται μια πιο συντονισμένη προσέγγιση και δεσμεύομαι να προσπαθήσω για κάτι τέτοιο μαζί με την Επίτροπο Ρέντινγκ και με άλλους ώστε η μετανάστευση, το άσυλο, οι εξωτερικές απειλές και το διασυνοριακό έγκλημα να ε, αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας εξέτασης. Πιστεύω ότι τα συστήματα που αναφέρατε μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Όπως είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, θα πρέπει καλύτερα να μπορούμε να ενώσουμε τις τελείες, διότι ε, απέτυχε και θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιες αποτυχίες στο μέλλον. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε αντί να δημιουργούμε νέα συστήματα πριν να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε. Όπως σας είπα, θέλω επισκόπηση της όλης αρχιτεκτονικής ε, που να λαμβάνει υπόψη όλα τα κριτήρια. Το κόστος, ε, την προστιθέμενη αξία, την αναλογικότητα, την προστασία των δεδομένων κλπ. Και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό προτού ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε νέα συστήματα. Και θα πρέπει το ΣΥΣ να αρχίσει να λειτουργεί πριν καν φτάσουμε στο σύστημα εισόδου-εξόδου. Πολύ καλά τα νέα αυτά. Υπάρχει άλλη πλευρά του θέματος, η έλλειψη επιχειρησιακής συνεργασίας. Ε, στις 9 Ιανουαρίου ε, στη Σλοβακία έγινε, τεστ, έγινε δοκιμή του αεροδρομίου. Ε, νέα, εννέα βόμβες τοποθετήθηκαν σε, σε βαλίτσες ταξιδιωτών ε, και μία βόμβα αυτή δεν εντοπίστηκε. Έφτασε στο Δουβλίνο όταν ε, ε, οι Ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν τις Σλοβάκικες, αυτές ε, δήλωσαν άγνοια και καθυστέρησε πολύ το θέμα. Αυτό είναι το τρομερό παράδειγμα και δείχνει το πραγματικό πρόβλημα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες και μεταξύ μας. Η συνεργασία των διαφόρων αρχών. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που αποσπούν την προσοχή μας από το βασικό θέμα, τη συνεργασία της αστυνομίας και ε, εντό των κρατών μελών, πόσο μάλλον ε, διασυνοριακά και ε, διατλαντικά. Ευχαριστώ. Αυτό είναι και φιλοσοφικό θέμα. Είμαστε άνθρωποι όλοι. εσεί αναφέρατε ένα παράδειγμα. Εγώ μπορώ να σα αναφέρω πολλά και από τη χώρα μου και από άλλε χώρε όπου οι αστυνομικέ αρχέ δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίε που ήταν διαθέσιμε. Και για το λόγο αυτό διαπράχθηκαν εγκλήματα, υπέφεραν άνθρωποι. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τελείω, ό,τι και να κάνουμε αλλά όπως είπατε θα πρέπει να μπορούμε καλύτερα να συνδυάζουμε τα μέσα που ήδη έχουμε, να δούμε πώς τα χρησιμοποιούμε, πώς τα αναλύουμε, πώς συνεργαζόμαστε, πώς οι υπηρεσίες μας γίνονται πιο αποτελεσματικές και πώς εμπιστευόμαστε ένα τον άλλον κατά την ανταλλαγή πληροφοριών. Και ελπίζω να μπορέσω να συμβάλλω σε αυτό. Αλλά άνθρωποι δουλεύουν με τα θέματα αυτά, πάντα θα γίνονται λάθη. Thank you. Mrs. Again. Κυρία Μπόσκουρ, ξανά ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας περιμένουμε η Κομισιόν να κάνει μια νέα πρόταση ε, κανονισμού για περιοριστικά μέτρα εναντίον ατόμων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλκάιδα, τον Σάμα Μπιν και τους Ταλιμπάν με, άρθρο, βάση το άρθρο 75 ε, της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια της, συνθήκης, στα πλαίσια της συναπόφασης. Αντίθετα, βασιστήκατε στο άρθρο 215 που ε, εξαιρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία. Δεσμεύεστε να σεβαστείτε τις ε, συνθήκες, ε, συνα... συγγνώμη, τις και τους όρους συναπόφασης με βάση το άρθρο 75 και ένα γενικό πλαίσιο για τα περιοριστικά μέτρα ανθρώπων αυτών, ε, παραδείγματο χάρη πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ούτω ώστε να αποφασίσουμε με βάση το άρθρο 75 και να υπάρχει και δημοκρατική, αν θέλετε, λογοδοσία. Ναι, θυμάμαι αυτή τη συζήτηση. Την κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια πριν από ένα μήνα. Ε, θυμάμαι ότι και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και της Κομισιόν ε, συμφώνησαν ότι το άρθρο 215 θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά το πάγωμα σε διεθνές επίπεδο ε, περιουσιακών στοιχείων ε, και δεν συμφωνήσαμε με την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά ε, το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 65. Αυτή είναι όμως μια διαμάχη, ας πούμε, μεταξύ των νομικών υπηρεσιών. Εγώ θέλω να είμαστε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοιχτοί και διαφανεί απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό είναι περισσότερο θέμα της συναδέλφου μου της κυρίας Άστον. Ε, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το άρθρο 215 θα πρέπει να εφαρμοστεί και όχι να χρησιμοποιηθεί και όχι το άρθρο 75. Ετοιμάζεστε, ε, να κάνετε μια πρόταση ε, για τα άτομα που δουν με αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το 75 στην απόφαση δηλαδή. Η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Και η δεύτερη. Είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε την πρότασή μας ε, στο ψήφισμα του περασμένου Δεκεμβρίου για να υπάρχει ένα δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ε, που θα προτείνουν στο Συμβούλιο τα πιο κατάλληλα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά μου φαίνεται καλή ιδέα να έχουμε αυτό το δίκτυο των εξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Ε, θα πρέπει να βλέπουμε και εκ του σύνεγγυς αλλά και με ανεξάρτητο μάτι ε, τι πρέπει να εφαρμόζουμε. Ε, θα πρέπει να είναι στοχευμένα αυτά τα περιοριστικά μέτρα και οι αθώοι να μην πέφτουν θύματα, να εστιάζουμε πραγματικά στους θύτες. Είναι λίγο ευρύ αυτό το εργαλείο, λίγο αμβλή, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για τον έλεγχο των πολιτών θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό και κατά πόσο σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Πάντως μου φαίνεται ως καλή ιδέα, μπορούμε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα που φίξατε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριο Στράσερ. Καλημέρα σας. Κύριε Μάστρον, Καλωσορίσατε θερμά τη νέα σας ιδιότητα εδώ. Επιτρέψτε μου εισαγωγικά να πω το εξής. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπει κανείς με ποιο δυναμισμό και πόση ενέργεια παρουσιάζεται εδώ την προσπάθειά σας και τη σχέδιά σας. Έρχομαι στην τρομοκρατία. Η τρομοκρατική απειλή ε, ήρθε ξανά παραμονές Χριστουγέννων στο προσκήνιο και συνειδητοποιήσαμε τι συμβαίνει με την αποτυχημένη τρομοκρατική απόπειρα. Αισθάνονται οι πολίτες να απειλούνται κυρίως από τον ε, Ισλαμικό εξτρεμισμό και τη τρομοκρατία που απορρέει από εκεί. Και αυτό θα πρέπει να βελτιωθούμε και στη συνεργασία μα. Γνωρίζουμε και το είπε ο ίδιο ο πρόεδρο Ομπάμα ότι αυτό δεν είναι τόσο θέμα έλλειψη πληροφοριών αλλά αξιολόγηση και επεξεργασία του. Και θέλω να επανέλθω και να σα παρακαλέσω να μα παρουσιάσετε τώρα μερικέ από τι προτάσει σα γενικά για τη στρατηγική ασφαλεία. Πού θέλετε να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσετε τα πράγματα για να έχετε καλύτερο συντονισμό, καλύτερη συνεργασία και με τους Αμερικανούς. Danke. Ευχαριστώ. Κυρία Μάνστρομ. Yes, thank you. As, you say. Ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς, στη παραμονή των Χριστουγέννων μας έδειξαν τα γεγονότα ότι παραμένει σημαντική απειλή η τρομοκρατία και δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε σε τέτοια θέματα. Για τη συλλογή των δεδομένων έχουμε μέτρα και εργαλεία και ε, εσωτερικά αλλά και συμφωνίες με τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικός εταίρος μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και χρειάζεται αναθεώρηση και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών συνεδριάζουν αύριο και μεθαύριο ε, με τον Επίτροπο Ρεν και την ε, Υπουργό Ναπολετάνου των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνεργαστούν, θα συζητήσουν για μέτρα συνεργασίας και πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στο μέλλον. Είναι πολύ καλό το γεγονό ότι θα έρθει στο Τολέδο Υπουργό Εσωτερική Ασφαλείας των ΗΠΑ για να συζητήσει ε, και άμεσα με του υπουργού. Βεβαίω χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και προθυμία των κρατών μελών. Η Europol κάνει καταπληκτική δουλειά, αλλά καμιά φορά τα κράτη-μέλη είναι απρόθυμα να μοιράζονται τις πληροφορίες που έχουμε. Θα πρέπει να ε, οικοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κυκλοφορούν οι πληροφορίες για να προλαμβάνονται οι τρομοκρατικές απειλές και άλλα εγκλήματα στο μέλλον. Για την εσωτερική στρατηγική ασφαλείας... Βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, το σχέδιο για προστασία κρίσιμων υποδομών προστασία συστημάτων πληροφορικής και πληροφοριών μας στο κυβερνό έγκλημα. Εκεί υπολοιπόμεθα και υστερούμε γιατί και εκεί υπάρχει νέος τρομοκρατίας και θα κάνω αντίστοιχες προτάσεις συγκεκριμένε. για τη στρατηγική αυτή εσωτερικη ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος, ε, η κυρία Χιμένες Πεσερίλ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ, κυρία Μάρστρομ, που σας ακούω εισαγωγικά να μιλάτε για τα θύματα της τρομοκρατίας, γιατί δυστυχώς γίνεται λόγος μόνο μετά από μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση. Παραμένει όμως η απειλή και ο καθένας μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να είναι θύμα της τρομοκρατίας. Συμφωνείτε κυρία Μάστρομ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι μέχρι στιγμή στην Ευρώπη δεν έχει γίνει το παραμικρό για να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε την ομοθεσία των κρατών μελών σε θέματα προστασίας των θυμάτων της τρομοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι το Δεκέμβρη στην τελευταία ολομέλεια ο κύριος Μπαρό δεσμεύτηκε σε αυτό που του είπα να υπάρξει ευρωπαϊκός χάρτης για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Εσείς αναλαμβάνετε αυτή τη δέσμευση από την πλευρά σας και τι θα κάνετε για να υπάρχει αυτός ο ευρωπαϊκός χάρτης των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Κύριε Μάστρο. Ναι, στα ισπανικά απαντά η υποψήφη. Πολύ σημαντικό. Εγώ έχω φίλο που στη Μαδρίτη πέθανε το 2004 στην Ατότσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και γνωρίζω ότι τα θύματα της τρομοκρατίας χρειάζονται περισσότερη προστασία και περισσότερη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε ορισμένα πράγματα. Υπάρχει ήδη ένα δίκτυο το οποίο συνδέει ε, για ανταλλαγή εμπειριών ε, τα διάφορα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Ε, υπάρχουν και πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση σωματείων συλλόγων, συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι πολύ καλό και μπορεί και πρέπει να επεκταθεί και να αναπτυχθεί. Ενδεχομένω στη στρατηγική ασφαλείας θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ε, ταμείο ασφαλείας έτσι ώστε να ε, προχωρούμε σε λήψη μέτρων για τα θύματα. Ε, θα μελετήσω τις υποσχέσεις που σας ε, έκανε και τη δεσμεύσεις του κυρίου Μπαρό για να έχουμε μία προσέγγιση αντίστοιχη στο μέλλον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Μακοβέη. Thank you. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 7-8 των πολιτών της ε, Ευρώπης θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στη χώρα τους, Συγγνώμη, 78% διορθώνει η ομιλήτρια. Συμφωνούν ότι η διαφθορά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στη χώρα τους και αναφέρομαι στα δεδομένα του Δεκεμβρίου του 2009 του Ευρωβαρόμετρου. Πρόκειται για πολύ πρόσφατα στοιχεία δηλαδή. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τα πρότυπα της ε, Διεθνούς Σύμβασης ε, κατά της ε, διαφθοράς, ε, με την επικύρωση της σύμβασης αυτής. Τι θα κάνετε για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή ε, μηχανισμού παρακολούθησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για αποτελεσματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Τι χρονοδιάγραμμα μπορούμε να αναμένουμε, ποια είναι τα μετρήσιμα στοιχεία που θέλετε, ποια είναι, ποιοι είναι οι αριθμητικοί στόχοι τους οποίους θέλετε να πετύχετε όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Ναι, η κυρία Μάρστρομ, ναι, ευχαριστώ. Ε, γνωρίζω την έκθεση αυτή, γνωρίζω και έκθεση της Greenpeace International που ε, μετράει τη διαφθορά σε όλες τις χώρες του κόσμου και με έκπληξη διαπίστωσα ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στον κατάλογο αυτό και μάλιστα σε πολύ χαμηλές θέσεις, κάτι που δεν είναι καθόλου καλό. Θα πρέπει λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι ε, στην διδασκαλία άλλων χωρών ε, σε θέματα καλής διακυβέρνησης ε, και διαφάνειας, θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς δουλειά στο δικό μας σπίτι. Στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης περιλαμβάνεται η ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Ε, θα υποβάλω ανακοίνωση σχετική. Είναι κάτι όμως που πρέπει να σκεφτούμε. Δεν λέω ότι είναι κακά αυτά που έχουμε, θα πρέπει όμως να δούμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα θέματα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Του χρόνου το Δεκέμβριο θα έχουμε μέρα, μια ημέρα κατά της διαφθοράς και στα πλαίσια αυτής πιστεύω θα μπορέσουμε να υποβάλουμε προτάσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά ε, την ε, διαφθορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωση, γιατί είναι σημαντικό το θέμα και είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα του πολίτε. Ευχαριστώ κυρία Μακομπέη. Ευχαριστώ. Μια διευκρίνηση. Η ερώτησή μου αναφερόταν ακριβώς στον, πρόγραμμα, στον μηχανισμό ε, παρακολούθησης ε, που αναφέρεται στο πρόγραμμα της στοχόρμης που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και επίσης πώς βλέπετε την εντολή σας στη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ε, σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, διότι η διαφθορά αφορά την απάτη. Ναι, φυσικά συνδέονται στενά τα δύο θέματα αυτά και πρόκειται για έργο του συνόλου της Κομισιόν να ε, διασφαλίσουμε αυτά που δίνουμε να είναι καθαρά. Ξέρετε, έχετε μεγάλη πείρα στο θέμα αυτό. Εσείς ε, γνωρίζετε πάντως ότι είναι ευθύνη του συνόλου του σώματος των ε, επιτρόπων και ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο έχει κάνει πολλά για να διασφαλίσει την ε, λογοδοσία σε θέματα που αποτελούν ευθύνη της Επιτροπής. Ξέρω επίσης ότι το Συμβούλιο εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό, όπως επίσης και εσείς, το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τον μηχανισμό παρακολούθησης, θα πρέπει να εκπονήσουμε κριτήρια μετρήσιμα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και επίσης να έχουμε ένα σύστημα ε, name and shame, όπου ονοματίζουμε και ντροπιάζουμε δηλαδή τους ε, παραβάτες. Ε, κάτι τέτοιο. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε. Θα υποβάλω πιο συγκεκριμένε προτάσεις, διότι συμφωνώ μαζί σα, ότι θα πρέπει να είναι απτό και συγκεκριμένο το πρόγραμμα αυτό, να μην είναι απλά ωραία λόγια. Το γνωρίζουμε αυτό. Ευχαριστώ κυρία Χέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σεσίλια, στην, ε, στις γραπτές σου απαντήσεις ε, είπες ότι ε, θα υποβάλεις πρόταση κατά της εμπορίας ανθρώπων φέτος. οι συνάδελφοί μου από την σοσιαλιστική ομάδα το επικροτούν αυτό, διότι πρέπει πράγματι να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Εσύ πώς βλέπεις τη δυνατότητες, τις δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη. Θα πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση υπηρεσιών από ανθρώπους ε, που έχουν πέσει θύματα Εμπορία ανθρώπων. Ε, ο Επίτροπος Παρό υπέβαλε προτάσεις. Ε, η Σουηδική Προεδρία όμως δεν κατάφερε να πετύχει συμφωνία στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Μάλστρομ. Ευχαριστώ όπως είπα και νωρίτερα. Πράγματι θα, υποβα... θα επανυποβάλλω την πρόταση αυτή. Πολύ κοντά βρεθήκαμε στην εξέβρεση συνένεση, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που άπτονται των ποινών ε, για τα οποία δεν επιτεύχθη συμφωνία. Θα επανυποβάλλω την πρόταση όμως ε, και ε, στα πλαίσια της ε, συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την ισχυρή αφοσίωση που υπάρχει εδώ στο Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση διότι είναι ένα τρομερό έγκλημα το οποίο διαπράτεται καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέοι άντρες, νέες γυναίκες πέφτουν θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Πράγματι είναι αλήθεια ότι η ζήτηση είναι σημαντικό πρόβλημα ε, στη Σουηδία έχουμε σχετική νομοθεσία που φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις για το θέμα αυτό και η Κομισιόν δεν έχει ε, αρμοδιότητα να εναρμονίσει το θέμα αυτό, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να συζητιέται συνέχεια το θέμα της ζήτησης όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων. Ε, σκοπός μου είναι να να υποβάλω την πρόταση και ελπίζω να περάσει. Ελπίζουμε στην ε, συμφωνία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ευχαριστώ η κυρία Χέτ πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αυτή. Μιλάμε πολύ για την ποινική πτυχή, ε, ποιες ποινές θα πρέπει να επιβάλλονται, αλλά για να προοδεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε και τα προληπτικά μέτρα καθώς και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ζήτησης όπως είπε. Ξέρουμε ότι σχεδόν το 80% ε, της, ε, του όγκου της εμπορίας ανθρώπων αφορά ε, σεξουαλική εκμετάλλευση. Θα πρέπει λοιπόν να θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπεις τη σχέση ανάμεσα στην πορνεία και την εμπορία ανθρώπων. Ναι, φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι που εντάσσεται σε διάφορες πολιτικές μας. Ε, θα πρέπει να ε, ενεργήσουμε προληπτικά. Είναι κάτι που είπα και στην κυρία Πάουερ, Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα θύματα Πιστεύω ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην πορνεία και στην εμπορία ανθρώπων, υπάρχει ζήτηση και έτσι ε, πραγματοποιείται το εμπόριο αυτό. Ε, αλλά όπως σας είπα, οι συνθήκες στα διάφορα είναι διαφορετικές. Ε, θα εξετάσουμε λοιπόν πρώτα την οδηγία αυτή. Θα συζητήσουμε και το θέμα της συζήτηση ε, αργότερα, αλλά δεν ε, υπάρχουν ε, ακόμα προβλέψεις για εναρμόνιση στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ Σεσίλια. Χαίρομαι πολύ που εσύ βρίσκεσαι εδώ μετά από τα πολλά χρόνια σου ε, ως Ευρωβουλευτής, ε, μετά από τις ώρες και μέρες που έχεις περάσει μαζί μας, ε, πιστεύω ότι ε, έχεις κερδίσει εμπιστοσύνη και στο σεβασμό των συναδέλφων σου. τώρα ακούμε τα σχέδια σου για... Τώρα ακούμε τη δέσμευσή σου να ασχοληθεί με τα θέματα πολιτικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. περιέγραψε σε συγκεκριμένα μέτρα. Χρειαζόμαστε όμως και ένα μακροπρόθεσμα όραμα. Πώς θα χειριστούμε την ανάγκη για ανθρώπινα δικαιώματα, ε, μια αλληλεγγύη στον τομέα της ε, μετανάστευσης. Ε, η κυβέρνησή μας έχει σύγχρονη νομοθεσία όσον αφορά την μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Θα ήθελα να μας παρουσιάσεις το όραμά σου για, το, ε, για τη μελλοντική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να παρουσιάσω το όραμά μου Φυσικά στον ιδανικό κόσμο δεν θα υπάρχουν σύνορα ε, και όλοι θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν έχουμε δημοκρατία και ε, υψηλό επίπεδο ανάπτυξη σε όλες τις χώρες. Και φυσικά από το στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να στηρίξει την δημοκρατία, την ευημερία σε όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν ε, ευνοεί την σταθερότητα στον ε, κόσμο όσο το να περάσουν τα δικτατορικά καθεστώτα σε δημοκρατικά. Δυστυχώς όμως δεν ζούμε σε ιδανικό κόσμο και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται στην ευθύνη, την προβλεψιμότητα, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Θέλω πολιτική ασύλου όπου να μπορούμε να προστατεύσουμε αυτού που το έχουν ανάγκη. Θα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι υπό ποιε συνθήκε θα του παρέχεται η προστασία αυτή. Θέλω πολιτική ε, που να, ώστε, να μπορούμε να δεχτούμε και νόμιμους μετανάστευσης και νόμους μετανάστες και θα πρέπει και αυτοί να ξέρουν υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είναι αυτό δυνατό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την λαθρομετανάστευση ε, Πολλοί μίλησαν για τις τρομερές συνέπειες της λαθρομετανάστευσης. Σε χιλιάδες πνίγονται στη Μεσόγειο κάθε χρόνο. Πολλοί πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ε, γίνονται σκλάβοι ε, ή ε, εργάζονται υπό καθεστώς εκμετάλλευσης σε όλο τον κόσμο. Και πρόκειται για ανθρώπους φτωχού, οι οποίοι θέλουν να ε, να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Δεν μπορούν να έρχονται όλοι αυτοί στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Θέλω αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο καθαρά ε, και με όσο γίνεται πιο ανθρώπινο τρόπο και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ κύριε Κορατσαμπίλτ. Ευχαριστώ Σεσίλια για την σαφή σου απάντηση. Τώρα θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Ε, σε πολλές από τις κοινωνίες μας ε, υπάρχουν ε, εξτρεμιστικές δυνάμεις οι οποίες αυξάνονται και που δεν συμμερίζονται τις ανθρωπιστικές μας αξίες. Θεωρούν ότι έχουμε υπερβολικά πολλούς μετανάστες και πολλοί φοβούνται ότι οι πολλοί μετανάστες θα απειλήσουν την ασφάλειά τους και τις δουλειές τους. Η οι πιο ευάλωτοι μετανάστες είναι τα ασυνόδευτα παιδιά. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορείς εσύ να κάνεις, ε, τι δέσμευση μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα για να αποφύγεις τα αθώα παιδιά αυτά να είναι ευάλωτα στη δική μας κοινωνία. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ανθρώπινη μεταχείρισή τους και τι μπορείς να κάνεις για να επανενώνονται με τις οικογένειές Ευχαριστώ Σεσίλια. Η κυρία Μάλστρομ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί σε ένα λεπτό. Το πρόβλημα με την ε, ε, ξενοφοβία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ε, ένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία, να συμβάλλουν και αυτοί στην κοινωνία. Όσον αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά, που είναι πρόσφυγες. Αυτό είναι αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός σε πολλές χώρες και σύντομα θα υποβάλω πρόταση για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στρατηγικά στον τομέα αυτό. Ε, τα συνόδευτα παιδιά φτάνουν ε, επειδή έχουν πέσει θύμα ε, εμπορίας ανθρώπων. Μερικά έρχονται μόνα τους και μερικά είναι παιδιά που ε, ε, νόμιμα έρχονται και έρχονται από διάφορες χώρες. Χρειαζόμαστε όμως μια κοινή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα δικαιώματα των παιδιών αυτών, το δικαίωμα επανένωσης με τις οικογένειές τους, ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα παιδιά. Θα πρέπει όμως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, διότι είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό στην Ευρώπη. Το φθινόπωρο θα υποβάλω σχετική πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Πορσελίνο. Κυρία Μάλστρομ, σήμερα μιλήσατε πολλές φορές για τη Λιβύα. Ε, μια χώρα που ακούστηκε σε μια κοινοβουλευτική συζήτηση ότι είναι μια ανεξέλεγκτη χώρα. Σήμερα μιλάμε για μια συμφωνία με αυτή τη χώρα που αφορά τη διαχείριση των συνόρων. Το άσυλο, ε, η λαθρομετανάστευση είναι θέματα που μας απασχολούν. Η Λιβύη όμως δεν, δεν, δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, τι δικαιώματα α, θα εξασφαλίσετε μάλλον ότι δεν θα υπάρξει επαναπροώθηση των ανθρώπων ε, προς τη Λιβύη. Πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Για το τελευταίο σας ερώτημα. Εγώ φυσικά θα έρθω στην Επιτροπή σας και θα σας ε, εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές προοδεύουν. Η πρόοδος είναι πολύ μικρή. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Ε, η Λιβύη όντω δεν έχει προσυπογράψει διεθνεί συμβάσει. Όμω έχει υπογράψει μια Αφρικανική σύμβαση για το πώ ε, πρέπει να μεταχειρίζονται οι χώρε αυτέ του ε, πρόσφυγε. Και είπαν ότι θέλουν να μεταφέρουν αυτά τα μέτρα στην εθνική του νομοθεσία. Αυτό είναι καλό το, το αντιμετωπίζουμε θετικά. Θέλουμε, λέμε στη Λιβύη, πώ να μα υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθειά, σε αυτή την προσπάθειά σας. Ε, αυτό του ρωτήσαμε από πλευρά Κομισιόν. Αλλά η Λιβύη δεν έχει απαντήσει, Επομένω είμαστε σε μια έτσι, κατάσταση αβεβαιότητα. Είναι μια σημαντική χώρα αυτή, σημαντικό γείτονα, σημαντική χώρα διέλευση, ε, χώρα από την οποία εκπορεύονται και μετανάστε και πρόσφυγε, αλλά θέλουμε η χώρα αυτή να σεβαστεί τι διεθνεί συμβάσει. Η Κομισιόν δίνει ήδη πολλά λεφτά στη Λιβύη και είναι διατεθειμένη να κάνει πολύ περισσότερα για να ενδυναμώσει τη Λιβύη, να δημιουργήσει θεσμούς, να οικοδομήσει το σύστημά τους. Ε, συνεργαζόμαστε πολύ με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες που δραστηριοποιείται στη Λιβύη. Βεβαίω ε, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ε, με τη Λιβύη, αλλά θέλουμε η Λιβύη να σέβεται τι διεθνεί τη υποχρεώσει. Ε, κυρία Μποσελίνο. Δεύτερη ερώτηση. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενημέρωση από πλευρά σας και αυτή η επαφή με το Κοινοβούλιο και αυτό το τονίζω. Θα ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση. Στις ε, γραπτές σας απαντήσεις δεν βρήκα καμία αναφορά για τους εποχικούς ε, εργαζόμενους. Σήμερα όμως μιλήσατε πολλές φορές. Τι προτάσεις θα παρουσιάσετε ε, ως Επίτροπος για αυτό το θέμα. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να τονίσω με αυτή την αφορμή για, κάτι, κάτι άλλο. Μιλήσαμε για την τρομοκρατία και για το οργανωμένο ε, έγκλημα, αλλά ποτέ δεν μιλήσατε για τη μαφία. Η μαφία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το οργανωμένο έγκλημα και σε όλα τα προβλήματα, την, τη διακίνηση, την ε, πορνεία, την εποχιακή εργασία, τα παιδιά, την σεξουαλική εκμετάλλευση. Σε όλα αυτά τα εγκλήματα η μαφία βάζει και αυτό το δαχτυλάκι της και όχι λίγο. Επομένως, πολύ συγκεκριμένα, για τη μαφία τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Κυρία Μάλστρομ. Yes, madam, thank you. On workers. Για τους εποχιακούς ε, εργαζομένους θα υποβάλω πρόταση. Για τα συνόδευτα παιδιά επίσης θα υποβάλω πρόταση για το πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό ε, με συντονισμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα στην Κοράτσα Μπίλτ, ε, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για τη μαφία τώρα. Ε, υπάρχει μια σημαντική διάσταση. Α, ο δάχτυλος της μαφίας δεν υπάρχει μόνο στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη. Και το ένα από τις μαφίες είναι στο οργανωμένο έγκλημα. Ε, το θέμα είναι πώ μπορούμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Μπαρό, ε, με την κυρία ε, Ρέντινγκ, συγγνώμη, και ο κύριος Μπαρό ασχολήθηκε με αυτό, ε, για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της μαφίας. αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν υπάρχει καταδίκη σε δικαστήριο. Η μαφία είναι θύμα του οργανωμένου εγκλήματος και πρέπει να ασχοληθούμε και συγκεκριμένα με τη μαφία. Επομένως θα την αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της εσωτερικής στρατηγικής ασφάλειας. Η κυρία Αλφάνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κυρία Μάλστρομ. Θα ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση για τη μαφία. Γιατί όπως είπε η κυρία Μπορσελίνο, σήμερα κανένας μίλησε για το πρόβλημα της μαφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατία. αλλά λίγα πράγματα έκανε για να μην πω τίποτα για τη μαφία. Κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από το οργανωμένο έγκλημα. Είναι ένα θέμα τελείως διαφορετικό αυτό τη μαφία. Ε, ξεκινάω με αυτή την προϋπόθεση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα καταρχά. και αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο που ε, στοιχείο και πρέπει να μα κάνει να σκεφτούμε. Η μαφία ε, υπάρχει και υπάρχει ως οικονομική παρουσία ε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για 250 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. 130 ε, από αυτά στην Ιταλία. αυτό είναι το οικονομικό προφίλ της Ιταλίας. η μαφία είναι το 8% του Ιταλικού ΑΕΠ. Τι πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι μπορείτε να προωθήσετε, νομοθετικές αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ. Κύριε Αλφάνο, δεν είμαι σε θέση να ποσοτικοποιήσω και να δώσω αριθμητικά στοιχεία ε, για την ε, δραστηριότητα της μαφίας. Αλλά ξέρω ότι όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και στον κόσμο ε, η μαφία ασχολείται με λαθρεμπορία ναρκωτικών, ε, διακίνηση ανθρώπων, παραχάραξη, απομιμήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας δώσω μόνο ένα νούμερο. Αν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ήταν μια χώρα, θα ήταν η 21η πιο πλούσια χώρα στην, στον κόσμο. Επομένως πολλά λεφτά είναι αυτά. Ε, δεν λέω ότι η μαφία ανακατεύεται σε όλα, αλλά... Αλλά ανακατεύεται σε πολλά. Και περιττώνει το λεφτό σε Ιταλό. Οι Ιταλικέ αρχέ εδώ και πολύ καιρό ασχολούνται με αυτό το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι και η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την ε, μαφία, γιατί επηρεάζει όλε μα τι κοινωνίε. Όπω είπα και στην κυρία Μπορσελίνο, στην εσωτερική στρατηγική, στρατηγική εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη μαφία. Να δούμε τι γίνεται με τι κατασχέσει. Φερρυπίν. Να προβούμε σε κατασχέσει. Η Ιταλία και πολλέ άλλε χώρε έχουν ε, μεγάλο απόθεμα έτσι, εμπειριών για την αντιμετώπιση τη Μαφία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ πιο ουσιαστικά για τη μαφία. Ευχαριστώ. Κύριε Αλφάνο, δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ. Δεν, ε, θα ήθελα να σας ε, αποσπάσω κάποιες ε, δεσμεύσεις. Να αναφέρω από αυτά που μας είπατε. Παραθέτω, είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρχών και μεταξύ των χωρών για το πρόβλημα της, του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι που λείπει κυρία Μάστρομ. Δεν υπάρχει ε, νομοθετική, αν θέλετε, συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Να σας ένα παράδειγμα που είναι ίσω το πιο γνωστό, αλλά και που δίνει ανάγλυφα το πρόβλημα. Θα θα θυμάστε την ε, σφαγή, τη μαφιόζικη σφαγή στη Γερμανία πριν από κάνα δύο χρόνια. Ένα ε, ένας εισαγγελέας Ιταλικός ζήτησε την κατάσχεση κάποιων περιουσιακών στοιχείων. Αλλά οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν γιατί δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία για τη μαφία. Έπειτα, μια και δεν υπάρχουν δεδομένα επίσημα. Δεν θα, δεν θα είχε νόημα να κάνουμε κάποιες μελέτες για να καταλάβουμε ε, την οικονομική σημασία της μαφίας. Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλές ανισότητες και διακρίσεις μεταξύ του πώς αντιμετωπίζουμε τα θύματα της μαφίας και της τρομοκρατίας. Στην Ιταλία υπάρχουν πάνω από 2.500 θύματα μαφίας. Ε, δεν είναι μικρό αυτό ο αριθμό. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην συνεχιστεί αυτή η διάκριση ανάμεσα στα θύματα τη τρομοκρατία και στα θύματα τη μαφία. Ε, είναι εξαιρετικά περίπλοκο αυτό το ζήτημα και δεν μπορώ να το απαντήσω σε ένα λεπτό. Φυσικά θα κοιτάξω τα νούμερα και τις στατιστικές που θα μου δώσετε και εσείς και οι συναδελφοί σας. Και φυσικά δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των θυμάτων. Τα θύματα βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος της Στοκχόλμης και είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει κοινή προσέγγιση για τα θύματα γενικά και ότι υπάρχει εγγύηση των δικαιωμάτων τους ε, στις διάφορες διαδικασίες. Βέβαια αυτή είναι ευθύνη της Επιτρόπου Ρέντινγκ, αλλά θα συνεργαστούμε για αυτό το θέμα. Ξέχασα την τελευταία σας ερώτηση. Ξέχασα κάποια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, μας επιτρέπετε να... λίγο χρόνο παραπάνω. Θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνδέεται με ένα θέμα που συζητήσαμε, που συζητάμε εδώ και δυόμιση ώρες, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους εγκληματίες και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Γιατί οι εγκληματίες περνάνε τα σύνορα. Άρα και εμείς θα πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητά μας να τους παρακολουθήσουμε, να τους ακολουθήσουμε. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών των διαφόρων χωρών. Ευχαριστώ κυρία Ρόιτοβα. Ε, ε, κυρία Μάλστρομ, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαι με την επιβολή ε, θεώρησης διαβατηρίου για τους Τσέχους πολίτες ο Καναδάς έδειξε ότι υπάρχουν ε, διάφορες κατηγορίες πολιτών της Ένωσης στα μάτια της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει απέναντι σε αυτή την πολιτική πραγματικότητα που είναι πάρα πολύ αρνητική. Τι προτίθεστε να κάνετε και μάλιστα ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να αποσύρει αυτές τις απαιτήσει θεώρησης ε, ο Καναδάς για τους Τσέχους πολίτες το συντομότερο παρακαλώ. Είστε διατεθειμένοι να θέσετε το θέμα αυτό ε, στα πλαίσια ε, των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνολική συμφωνία εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας με τον Καναδά. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρστον. Ναι, ευχαριστώ. Βεβαίως γνωρίζω το πρόβλημα αυτό και κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας το συζητήσαμε πολύ. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει πάρα πολύ σε εντατικότατες επαφές και συζητήσεις με τις καναδικές αρχές. Δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα, πάντως ε, υπάρχει πρόοδος και από την πρώτη μέρα θα αναλάβω το θέμα αυτό από τον Επίτροπο Μπαρό και άλλους επιτρόπους που ενέχονται για να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε για να βρεθεί λύση. Ευχαριστώ και πάλι. Η κυρία Ρόιτοβα. Είστε πρόθυμοι να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την αλληλεγγύη και να εγκρίνουν κοινά μέτρα. Again. Ε, δεν κατάλαβα, συγγνώμη την ερώτηση. Τι θέλετε να... μπορείτε να αναγκάσετε τα κράτη-μέλη να έχουν αλληλεγγύη με την τσεχική δημοκρατία στο θέμα αυτό και να εγκρίνουν κάποια κοινά μέτρα και θέματα αμοιβαιότητας δηλαδή. Βεβαίως και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσαν ότι έχουμε κοινή πολιτική εδώ και είναι πλήρης αλληλεγγύη με την τσεχική δημοκρατία απέναντι με τον Καναδά και εξηγούμε στις καναδικές αρχές ότι δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο την τσεχική δημοκρατία, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Έχουμε κοινή προσέγγιση εδώ και σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα, που νομίζω ότι θα λυθεί, θα έχουμε και κοινή απόκριση τα 27 κράτη-μέλη προς τον Καναδά. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα βρεθεί λύση. Είμαι αισιόδοξη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριο παπα Παπα-Νικολάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mr. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θα επανέλθω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Αναφέρθηκε ήδη και από εσάς και από συναδέλφους ότι τα μεγάλα κύματα λαθρομεταναστών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβαρύνουν δυσανάλογα κυρίως τα κράτη-μέλη της Νότιας Ευρώπης. Και συχνά αναφερόμαστε στην αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουμε ε, για την αντιμετώπιση της ροής λαθρομεταναστών και αυτό είναι αυτονόητο γιατί αυτοί που μπαίνουν στο νότο πολλοί από αυτούς κατευθύνονται προς το βορρά στην πράξη όμως έχουμε δει και αυτή είναι η πραγματικότητα ελάχιστη ουσιαστική πρόοδο στην επίδειξη της αλληλεγγύης. Σας ρωτώ λοιπόν και παρακαλώ για συγκεκριμένες απαντήσεις. Πώς σκοπεύετε με συγκεκριμένα μέτρα να κάνετε την αλληλεγγύη να δουλέψει στην πράξη. Και δεύτερον, πώς αντιλαμβάνεστε την επίδειξη αλληλεγγύης. Την αντιλαμβάνεστε σε εθελοντική βάση ή σε υποχρεωτική βάση μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Φυσικά γνωρίζω την πίεση που ασκείται σε κάποια κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ε, σε συγκεκριμένες εποχές. Και αυτό μας δυσκολεύει, ωστόσο η πλειοψηφία των μεταναστών, ε, λαθρομεταναστών και νομιμών έρχονται ε, από, με άλλους τρόπους, έρχονται αεροπορικά ή, με άλλους τρόπους. Ε, και όπως είπε ο κύριος Πουζετήλ και άλλοι, το πρόβλημα στη Μεσόγειο είναι ότι δημιουργούνται πολλές ανθρώπινες τραγωδίες και αποτελεί ευθύνη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά όσον αφορά την ε, αλληλεγγύη. Έχουμε μηχανισμούς, έχω δεσμευτεί να ε, ενισχύσω κάποιους από αυτούς, όπως είναι το Frontex. Θέλω να συνεργαστώ ε, με το πρόγραμμα της Μάλτας για να γίνει αυτό πιο μόνιμο κομμάτι της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επανεισδοχή, την επανεγκατάσταση. Ε, θέλουμε να πείσουμε τις χώρες να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό και άλλα. Και νομίζω ότι το σύστημα υποστήριξης ασύλου θα, το γραφείο υποστήριξης ασύλου θα βοηθήσει πολύ και δεσμεύομαι να το κάνω αυτό και με γειτονικέ χώρες, ε, να τις πείσω να συμμετάσχουν όσον αφορά την επανεισδοχή και να μας βοηθήσουν να προλάβουμε την ε, μετανάστευση. Ε, θα πρέπει φυσικά να δούμε το θέμα σφαιρικά, θα πρέπει να δούμε τις ε, διαφορές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες όσον αφορά την ευημερία και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Πολιτικά δεν είναι δυνατόν να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη. Μπορούμε να ενισχύσουμε τα μέσα, τα κίνητρα, μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική πίεση, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε υποχρεωτικό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Έχουμε οικονομικά και πολιτικά μέσα για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Θα τα χρησιμοποιήσω όσο γίνεται, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Σε συνεργασία όμως με το Κοινοβούλιο, η ε, Κομισιόν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη και να τους ζητήσει να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου πάλι. Αυτό που είπατε κυρία Υποψήφια Επίτροπε, να υπενθυμίσω κάτι που είδα στις αναλύσεις. Το 2008 το 25% από το σύνολο των λαθρομεταναστών που συνελήφθησαν, το 25% των συλλήψεων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, το 16% αν θυμάμαι καλά στην Ισπανία, το 15% στην Ιταλία και κάπου εκεί κοντά είναι και η Πορτογαλία. Ε, πώς σκοπεύετε για να δώσω έμφαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, με ποιο τρόπο και συνεχίζοντας σκοπεύετε να συνεισφέρετε στη δημιουργία νέων υποδομών υποδοχής για τους παράνομους μετανάστες και τους ετούντες άσυλο καθώς βεβαίως και στη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών με τέτοιο τρόπο που από τη μία να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για αυτούς και από την άλλη να εκφράζεται όσο πιο έμπρακτα γίνεται ε, η αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη ιδίω επαναλαμβάνω τη Νότια Ευρώπη, που δέχονται μεγάλα κύματα παράνομων μεταναστών. Ευχαριστώ, κύριε Μάνσομ. Ναι, πιστεύω ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αλληλεγγύης στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βοηθούν άλλα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη να ενισχύσουν τις δυνατότητες ε, υποδοχής που έχουν με μεταφορά τεχνολογίας, ε, εμπειρογνωμοσύνης, εμπειριών Υπάρχουν όμως και οικονομικοί πόροι που μπορούν να βοηθήσουν. Οι χώρες που υφίστανται τεράστιες πιέσεις, είτε προσωρινά είτε πιο μόνιμα, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται κόσμο. Αυτό συνεχίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη λειτουργεί, μπορεί να ενισχυθεί πιστεύω και είναι καλός τρόπος να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Έχει πολλές διαστάσεις η αλληλεγγύη. και θα πρέπει να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, αλλά να μην δυσμονούμε ποτέ ότι έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε εκείνους που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε υποδομές υποδοχής. Και θα κάνω προτάσεις, θα προσπαθήσω τουλάχιστον για να εναρμονίσουμε αυτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία Μάλστρομ, ενδιαφέρουσες ώρες περνάμε, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων και την αρχή της ε, αναλογικότητας την ε, πολιτική ασφαλείας. Όλα αυτά εγώ τα καλωσορίζω και χαίρομαι που τα λέτε, αλλά δεν ξέρω ότι πρεσβεύεται σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό έχω να σας κάνω ερωτήσεις λεπτομέρειες. Η απάντηση θα είναι ναι ή όχι. Πρώτον, θα αναθεωρήσετε την δυσανάλογη οδηγία προφανώς για τη ε, διατήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, δικαίωματα των πολιτών για το φάκελό τους, για τα στοιχεία που συλλέγονται σε ό,τι αφορά την αστυνομική, τη δικαστική συνεργασία και ε, τις εποπτικές αρχές. Και τρίτη ερώτηση. Θα προτείνετε πλήρη αποζημίωση σύμφωνα με την ΕΣΔΑ ε, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν πρόκειται για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες μη κοινωτικές χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάσο. Θα μπορούσα να απαντήσω καταφατικά και στι τρει ερωτήσει, αλλά χρειάζεται λεπτομερής απάντηση και κάποιε αποχρώσεις. Η οδηγία για τη φύλαξη των προσωπικών δεδομένων θα αναφερθεί του χρόνου. Θα γίνει μια αξιολόγηση και βεβαίω θα δούμε όλα αυτά τα θέματα ε, την προστασία των δεδομένων, την αναλογικότητα, το κόστος, τη χρησιμότητα, τη σκοπιμότητα. Την πλήρη αποζημίωση βεβαίω είναι ένα θέμα που είναι στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι πολίτες των κρατών μελών εντάσσονται στην προστασία μας και διέπονται από τις αρχές μας και θέλουμε να τις προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς. Υπάρχει η ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και είναι ένα θέμα στο οποίο σίγουρα αναφέρθηκε και η κυρία Ρέντινγκ. Και ένα στοιχείο της αναθεώρησης του συστήματος δεδομένων και του διαρκούς διαλόγου που πρέπει να έχουμε και με τις εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές είναι πώς μπορεί να έχει πληροφορίες ο πολίτης σχετικά με τα στοιχεία που συλλέγονται για τον ίδιο και κατά πόσο αυτά διαβιβάζονται σε άλλους. Αυτό μπορεί να είναι εις βάρος του να επηρεάζει αρνητικά τη ζωή του. Αυτό διαφέρει από σύστημα συλλογή σε σύστημα συλλογή, αλλά θα συνεργαστώ με την κυρία Ρέντινγκ και για αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσω. Ο κύριο Άλμπρεχτ για σημαντική ερώτηση. Δεν ξέρω τελικά αν ήταν ή όχι αυτό που απαντήσατε. πάση περιπτώσει. Για τα μέτρα ασφαλείας Συχνά γίνεται λόγος για γεγονότα και πληροφορίες υποτιθέμενες που ε, αποδεικνύουν ότι χρειάζονται αυτά τα μέτρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους καλούνται κάποιοι πάνω. Δεν παίρνουμε αυτά τα στοιχεία. Ας πούμε η κυρία Αναπολιτάνο, στην ίδια επιτροπή, η Αμερικανίδα υπουργό είπε ότι δεν είναι περιοριστική όρια από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα με τη συνθήκη έχουμε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα στα έγγραφα σε όλα τα στάδια εκπόνησής του. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα μας στέλνετε όλα τα έγγραφα αμέσω, κυρία Μάλστρομ. Όχι. Διότι δεν μπορώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Είναι περίπλοκα θέματα και σημαντικά. Εγώ δεσμεύομαι να βεβαιωθώ ότι εσείς ως συνομοθέτης θα έχετε την ίδια πληροφόρηση για όλα τα θέματα, για όλες τις προτάσεις με το Συμβούλιο. Ναι, γνωρίζουμε ότι σε θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης υπάρχουν και έγγραφα διαφαθμισμένα. Ορισμένα δίνονται με διαφορετικούς τρόπους στον πρόεδρο, στον συντονιστή, στους συντονιστές, στους ηγητές και χωρίς να είναι δημόσια. Αυτό θα συζητηθεί στη νέα ε, απόφαση πλαίσιο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι ο κύριος Μπαρόσο είναι ιδιαίτερα προσιλωμένος σε αυτό και θα το συζητήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των εμπιστευτικών εγγράφων ε, παντού για τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι θα επανέλθει πολύ σύντομα ο κύριο Μπαρόσο. Ίσως και στην ίδια την ομιλία που θα εκφωνεί στο Κοινοβούλιο όταν θα ψηφίσετε για την Επιτροπή. Εγώ πάντως δεσμεύομαι ότι θα έχετε όσο γίνεται περισσότερη πληροφόρηση και ίση ε, με το Συμβούλιο όταν συνομοθετείτε. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Φαχών. Thank Ξέρω ότι όλοι είμαστε κουρασμένοι. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, ιδίως για αυτούς που δεν είναι τμήμα κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Μιλάει για τους πολίτες της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας, οι οποίοι περιμένουν σε ατελείωτες ουρές μπροστά στις πρεσβείες για να πάρουν θεωρήσεις για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τραγικές ιστορίες, ειδικότερα για τους πιο νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει όπως έδρασε και στην περίπτωση της Βοσνία, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου και θα προτείνει την κατάργηση των θεωρήσεων, παρότι δεν έχουν ακόμα, δεν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Ε, θα πρέπει ε, είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε για την Αλβανία και τη Βοσνία ζηγοβίνη την απελευθέρωση την υποχρέωση των θεωρήσεων πριν τις διακοπές, τις καλοκαιρινές, τον Ιούλιο ας πούμε. Ε, πότε θα πέσουν όλοι οι τύχοι για τις ε, θεωρήσεις και για το κοσφοπέδιο. Η διευκόλυνση των θεωρήσεων είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο και αισθάνομαι τιμή που ήμουν τμήμα της σπουδικής ε, ομάδας για να δώσουμε αυτή τη διευκόλυνση στη Μακεδονία και στη Βοσνία. Ε, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε κυρία Φαχών, για τους νέους, γιατί έτσι θα σανθρώ την τμήμα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία, θα πρέπει επίσης όπως και για την ε, διεύρυνση, να έχουμε και εδώ κάποια κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται. Υπάρχουν για τις, ε, όταν υπάρχουν και για τις τρεις χώρες, θα προχωρήσουμε. Για την ε, Αλβανία και τη Βοσνία Ερσεγοβίνη ακόμα δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί και εγώ δεσμεύομαι να βοηθήσω και να υποστηρίξω αυτές τις χώρες στο ταξίδι αυτό μέχρι να φτάσουν ε, στην πόρτα της εισόδου που θα πέσουν αυτά τα τείχη. Η Κομισιόν μπορεί να τι βοηθήσει, αλλά και αυτές πρέπει να κάνουν την προσπάθειά τους. Πότε ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια, πότε τελειώνει αυτή η προσπάθεια. Δεν μπορώ να δώσω μια ημερομηνία εγώ γι' αυτό. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα από πλευρά του. Και ελπίζω ε, να συμφωνήσουμε κατά τη διάρκεια του 2010. Αλλά αυτό εξαρτάται από τα κριτήρια. Το κοσυφοπαίδιο δεν ήταν τμήμα ε, του διαλόγου για τις θεωρήσεις από την αρχή. Αλλά η Κομισιόν και ο προκάτοχό μου, ο κύριο Παρό, δεσμεύτηκε προσωπικά να συνεργαστεί με το Κοσμοπέδιο για να δει τι μέσα διευκόλυνση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα επανέλθω λοιπόν ενώπιον του Κοινοβουλίου να σα ενημερώσω για αυτό το θέμα. Η κυρία Φαχών ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι η Βοσνία, η Ζεγοβίνη και η Αλβανία πρέπει να εκπληρώσουν όλες τις προϋποθέσεις όπως και άλλες χώρες έκαναν, ε, έκαναν προσπαθειά τους. Αλλά πέρυσι τον Ιούλιο η Σερβία και το Μαυροβούνιο δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια και όμως η Κομισιόν πρότεινε να υπάρξει αυτό το καθεστώς απελευθέρωση των θεωρήσεων. Η Βοσνία, η Ζεγοβίνη και η Αλβανία αποκλείστηκαν όμως από την προσπάθεια. Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και για αυτές τις δύο χώρες, να γίνει μια σύσταση δηλαδή στις αρχές της Άνοιξης. Και μια συμπληρωματική ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την, τα ταξίδια των Ευρωπαίων πολιτών ε, στις ε, ΗΠΑ, θα πρέπει να καταβληθούν κάποια τέλη, κάποιες πληρωμές πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν οι πολίτες μας να μεταβούν στις ΗΠΑ. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, για το πρώτο ερώτημα. Βεβαίω, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Βοσνία, ε, Ζεγοβίνη και την Αλβανία για να εκπληρώσουν αυτά τα κριτήρια. Η Κομισιόν τελικά, όταν πιστέψουν ότι, πιστέψει ότι είναι έτοιμε αυτέ οι χώρε, θα κάνουν την πρόταση. Αλλά οι υπουργοί θα πάρουν την απόφαση. Και ξέρετε πολύ καλά, επειδή είναι υπουργοί εξωτερικών, δεν είναι πάντα πρόθυμοι να πάρουν αυτή την απόφαση. Ε, θα προωθήσουμε την ίση μεταχείριση, αλλά πρέπει να εκπληρώσουν τα κριτήρια και τι προποθέσει για τη δεύτερη ερώτηση. Θα το εξετάσουμε το θέμα και έχουμε πει στις αρμανικανικές αρχές ότι αν το έστα αυτό σημαίνει, σημαίνει θεώρηση, σημαίνει βίζα τελικά, αν είναι ένα επιπρόσθετο τέλος, ε, τελικά διαφωνούμε ε, στεναρά. Το εξετάζει το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή και περιμένουμε κάποια στιγμή να έχουμε απάντηση. Αλλά το παρακολουθούμε εκ του και είχαμε πει ξεκάθαρα στι αμερικανικές αρχές τι πιστεύουμε για αυτό το τέλος. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία υποψήφια, σήμερα ακούσαμε πολλά ε, και είπαμε πολλά για δικαιώματα, δικαιώματα μειονοτήτων, για βοήθεια των παιδιών, όλα σημαντικά είναι και μας συγκινούν. Αλλά σε όλα αυτά τα θέματα έχουμε μια ειδική νέα επίτροπος που είναι αρμόδια και ονομάζεται κυρία Βιβιάννα Ρέντινγκ που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Τέτοιο χαρτοφυλάκιο εσείς στο μέλλον είστε το πρόσωπο για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης και ελπίζω να έχετε και επίγνωση του γεγονότος ότι αυτό είναι πρώτη σας προτεραιότητα. Θα ήθελα να γίνω και πιο συγκεκριμένος, γιατί πολλοί έχουν την αίσθηση ότι είχατε μια συμπαθή παρουσία εδώ, αλλά σε συγκεκριμένες δηλώσεις δυστυχώς κάπου δεν εμβαθύνατε. Παράδειγμα, ε, ρώτησαν οι φιλελεύθεροι και η συνάδελφος Αλφάνο για τη μαφία και μας απαντήσατε ότι ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ότι οι Ιταλικές αρχές θα το αντιμετωπίσουν. Ε, για μένα είναι αλλιώ η απάντηση. Άλλη ερώτηση τη κυρία Λάτφορτ και ρώτησε για την αντιτρομοκρατική ε, προσπάθεια για το, τη δικτύωση στην Ευρώπη. Είπατε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά πρόταση για δικτύωση των αρχών όχι. Γι' αυτό παρακαλώ, ε, απαντήστε μου συγκεκριμένα σε δύο-τρεις ε, υποθέσεις. Πρώτον, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Θα κάνετε πρόταση οδηγίας για τη δικτύωση των αρμοδίων διοκτικών αρχών στην Ευρώπη με τρόπο επιχειρησιακό όμως. Δεύτερον, Eurodac. Θα ήθελα να δεσμευτείτε ότι στα στοιχεία με τα δακτυλικά αποτυπώματα θα υπάρχει πρόσβαση σε αρχές ασφαλείας στην Ευρώπη. Και το τρίτο έχει να κάνει με το Frontex. Θα παρακαλούσα στο μέλλον να μας πείτε τι θα κάνετε όταν θα αναθεωρηθούν οι αρμοδιότητες του, θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν τις προδιαγραφές στα εξωτερικά σύνορα ανεξάρτητα. Αυτό τον καιρό δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν επιτρέπονται. Συγκεκριμένη απάντηση θέλω, ναι ή ου. Παρακαλώ, η κυρία Μάλμστρομ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Πρώτον, δεν είναι αντίφαση το να υπερασπίζεσαι τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Χέρι-χέρι πηγαίνουν. Δεν είναι ότι εγώ είμαι αστυνομία και η κυρία Ρέντινγκ ε, η καλή. Θα συνεργαστούμε για να υπερασπιστούμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων. Για το άλλο κύριε Βέμπερ που με ρωτήσετε, λυπάμαι, αλλά ένα μήνα είχα μόνο για να μελετήσω αυτό το τεράστιο ζήτημα. Ε, βρήθη πολλών θεμάτων πάρα πολύ ενδιαφερόντων αλλά και ε, περιπλόκων δεν μπορώ να σας απαντήσω πλήρως για όλα αυτά τα θέματα πριν αναλάβω. Αυτό ισχύει για όλους τους επιτρόπους, όλες τις επιτροπές. Δεν μπορούν να απαντήσουν σε όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ δεν γνωρίζω αρκετά τα πράγματα. Και εγώ θέλω να δεσμευτώ ότι οι προτάσεις που θα κάνω θα είναι θεμελιωμένες, στοιχειοθετημένες ε, με ε, αξιολόγηση και εκτίμηση. ήταν πάρα πολύ ανεύθυνο και επιπόλαιο να έρθω εδώ να σας απαντήσω πριν έχω μελετήσει σε βάθος όλα τα θέματα. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Και Νομίζω ότι απάντησα. Δεν ξέρω αν ήταν πρόβλημα διερμηνία. Δεν είπα εγώ ότι η μαφία ήταν μεγάλο Ιταλικό και μόνο πρόβλημα. Είπα ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους Ιταλούς διότι η μαφία είναι διάχυτη, έχει απλώσει τα πλοκάμια της στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Και ευρωπαϊκό βεβαίως πρόβλημα είναι και θέλω να έχουμε αντιμετώπιση ευρωπαϊκή, θα επανέλθουμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Βεβαίω βασιζόμενοι στην Ιταλική εμπειρία, γιατί οι Ιταλοί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από του άλλου. σω εγώ τα είπα με τρόπο ασαφή, δεν ξέρω. Ε, για το Eurodac, ναι, νέα πρόταση θα σα καταθέσω, με μια πρόταση στα πλαίσια τη Λισαβόνα πλέον και θα το συζητήσουμε. Το είπε και το Συμβούλιο, άλλωστε και δήλωσε ότι ε, θέματα ποινικού δικαίου θα πρέπει να ενταχθούν ε, πάντα στα πλαίσια της συνδέξης Λισαβόνας θα επανέλθουμε. Για τον οργανισμό Frontex αν κατάλαβα καλά, με ρωτάτε θα πρέπει να έχει εντολή για να θέτει κάποιες προδιαγραφές για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ναι, ναι, νομίζω, ναι, να έχουμε μια ενιαία τυποποιημένη διαδικασία με εκπαίδευση, με πραγματογνωμοσύνη, με γνώση, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη έχουν ένα κοινό επίπεδο και προδιαγραφές και πρότυπα φύλαξη των συνόρων. Ελπίζω να ήμουν αρκετά πλήρης και στα άλλα θέματα θα επανέλθω όταν θα τα έχω μελετήσει σε περισσότερο βάθος. Ευχαριστώ κύριος Βέμπερ, συμπροματική ευχαριστώ. Όλοι θέλουν να βάλουν τα θέματα ε, αυτά στη συζήτηση και βέβαια καλή επίτροπος θα είστε, δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να είστε και φιλόδοξοι επίτροπος για τα εσωτερικά θέματα και την ασφάλεια. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο σας, γι' αυτό θέλω φιλόδοξη υποψήφια με φιλόδοξη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, ήταν συγκεκριμένες. Ε, άκουσα για την αστυνομική συνεργασία ότι θα κάνετε συγκεκριμένη πρόταση και για την καταπολέμηση της μαφίας, για την παρακολούθηση και τη συνέχεια των προσπαθειών και για το Frontex ότι θα κάνετε την αξιολόγηση, αν φέρετε όλα αυτά τα συγκεκριμένα, τότε ελπίζω να είστε δραστήρια και φιλόδοξοι επίτροπος και στο μέλλον και χαίρομαι αν συνεχίσετε με αυτή σας τη φιλοδοξία. Mrs. Malmström, your turn, final turn, last Thank you. Τελευταία απάντηση. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια κύριε Βέμπερ. Αν διαβάσετε τα πρακτικά των, της ακρόασης, οι περισσότερες ερωτήσεις που μου κάνανε ήταν για το άσυλο και τη μετανάστευση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάστηκε και εγώ να μιλήσω περισσότερο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Αλλά μην ε, σας διαβεβαιώ ότι για την εσωτερική στρατηγική ασφάλειας δίνω μεγάλη σημασία και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο, θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, τις ε, οδηγίες τους οργανισμούς, τα agencies, για να καταπολεμήσουμε το διασυνοριακό έγκλημα, την τρομοκρατία, τη διακίνηση, το κυβερνοέγκλημα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να με απασχολήσει. Το έγκλημα που συνδέεται με τη μαφία κτλ. Θα κάνουμε προτάσεις, θα κάνω προτάσεις. Ε, έχω δεσμευτεί γι' αυτό. Όπως είπατε κι εσείς, Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, ελπίζω να τα ξαναπούμε και να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα ε, μπαίνοντα σε περισσότερε λεπτομέρειε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μάλστρομ, σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις. Ήταν μια μακρά ακρόση, ε, ήταν εξαντλητική η εξέταση αυτή, ήταν σκληρή αυτή η προσπάθεια εδώ και τρει ώρες τελειώσαμε την ώρα που είχαμε προαναγγείλει και τώρα για να αξιολογήσουμε την ακρόαση αυτή θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών σε αυτήν εδώ την αίθουσα στη 1.30 η ώρα. 1.30 ώρα το απόγευμα. Και μισή ώρα αργότερα, στις δύο η ώρα το απόγευμα, ε, θα συναντηθεί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην ίδια αυτή αίθουσα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Ε, κυρία Μάλστρομ και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και περιμένουμε με ανυπομονησία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.